Και έτσι καλωσορίζω τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, κύριο Ρέντσι. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε Σούλτς, κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τα λόγια που και εσείς απευθύνατε κύριε Πρόεδρε στο σώμα με αφορμή όσα συνέβησαν πριν από 70 χρόνια στο Auschwitz. Επιβεβαιώνω τη δέσμευση της κυβέρνησης και του λαού της Ιταλίας για τον αγώνα κατά αυτού του όνειδους που χαρακτήρισε την Ευρώπη και επί δεκαετίες ακόμα είναι κάτι που το θυμόμαστε όλοι. Έχουμε χρέος από το παρελθόν και πρέπει να κάνουμε μια επένδυση σοβαρή για τις μελλοντικέ γενιές. Ο χαιρετισμό σας, η ομιλία σας πρόεδρε, μας επιτρέπουν να μπούμε στην ουσία της ανασκόπησης του εξαμήνου της Ιταλικής Προεδρίας και να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε. Αφορμή είναι ο χαρακτήρας του τηλεμάχου, για να θυμηθούμε και την ελληνική μυθολογία. Ας σκεφτούμε αν σήμερα αυτά τα θεσμικά όργανα, αυτοί οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες που γνωρίζουμε, αυτοί οι εκπρόσωποι των περιοχών που σχηματίζουν το μεγάλο όνειρο της Ευρώπης, είναι σε θέση να αναλάβουν και να είναι άξιοι κληρονόμοι. Τι θα πει κληρονόμοι όμως. Για μας Ευρώπη δεν είναι απλώς η μνήμη, είναι η ελπίδα πάνω απ' όλα. Κοιτάζουμε στο μέλλον, όχι μόνο στο παρελθόν. Έχει τη θέρμη και το χρώμα της ευκαιρίας. Ευκαιρίας που θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο από την ανησυχία. Αυτούς τους έξι μήνες λοιπόν βρεθήκαμε στο ύψος των προσδοκιών αυτής της πρόκλησης. Οπωσδήποτε γνωρίζω ότι ο τύπος πριν περάσουμε σε αυτό το μεγάλο θύμα, θέμα, θα δώσουν ε, ε, έμφαση στα αποτελέσματα. Πες μας αν είσαι ικανοποιημένος στο τι έκανε για την Ευρώπη η Ιταλία. Είναι κακό ερώτημα αυτό, είναι κακή αρχή. Διότι στην πολιτική κανείς δεν είναι ποτέ πλήρως ικανοποιημένος. Αν είναι πλήρως ικανοποιημένος, καλό είναι να αλλάξει δουλειά δεν σκέφτεται κανείς ε, το ε, εξάμεινο μιας προεδρίας με γνώμονα το συμφέρον της ίδιας του της χώρας, αλλά με γνώμονα το πώς η Ευρώπη μπορεί να έχει ευκαιρίες για το μέλλον. Εμείς, οι Ιταλοί, οποιοδήποτε πολιτικού χρωματισμού, γνωρίζουμε τέλεια ότι η πρόκληση δεν αφορά τα του οίκου δεν αφορά μόνο το να παραμείνουμε στα στερεότυπα των ε, διαφορετικών μεταρρυθμίσεων σημαίνει ότι αν θέλει να παραμείνει πρωταγωνίστρια στο διεθνή ανταγωνισμό η Ιταλία πρέπει να αλλάξει. Και αυτούς τους έξι μήνες κάναμε πολλά. Κάναμε πολλά στη χώρα μας. Αυτά που εξυπηρετούν την Ιταλία λοιπόν τα αναλαμβάνουν οι Ιταλοί πολίτες, όχι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι Ιταλοί πολίτες γνωρίζουν πλήρως ότι τα τελευταία χρόνια φροντίσαμε να δώσουμε στην Ευρώπη πολύ περισσότερους πόρους από ό,τι πήραμε εμείς. Κάθε χρόνο η Ιταλία δίνει περίπου 20 δις ευρώ προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και παίρνει πίσω λιγότερο από το μισό. Αυτά τα χρόνια η Ιταλία συνέδραμε στην διάσωση χωρών φίλων αλλά και τραπεζικά ιδρύματα άλλων χωρών. Και όχι από γενεοδορία, αλλά γιατί πραγματικά έχει βαθιά πίστη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. δεν ε, πήραμε ούτε ένα ε, λεπτό ευρώ από ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να σώσουμε τα δικά μας τραπεζικά ιδρύματα. Όχι. Για την Ευρώπη έγιναν όλα αυτά. Πιστεύουμε στην Ευρώπη. Και δεν ερχόμαστε ως Ιταλία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να ζητήσουμε βοήθεια. Άτι, αλλά για να προσφέρουμε τη μεγάλη μας ιστορία που ξεκίνησε στη Ρώμη με την υπογραφή της συνθήκης. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε και πολύ νωρίτερα θεμελιώνεται στις αξίες που έκαναν μεγάλη τη χώρα μας και μεγάλη την Ήπειρό μας. Αυτή είναι η δική μας ιδέα για την Ευρώπη. Ένας τόπος ελπίδας για τις μελλοντικέ γενές. Και ξέρουμε ότι τα δικά μας προβλήματα πρέπει να τα, να λύσουμε ε, στο δικό μας, στη δική μας χώρα, όπως με το Σύνταγμα, με τη δικαιοσύνη, με τη δημόσια δίκηση, όλες τις πραγματικότητες που απασχόλησαν την Ιταλική Βουλή αυτό το εξάμεινο κίνητρό μας για το ε, τελικό εξάμεινο ήταν η ευρωπαϊκή μας πρόπτικη που είναι τόσο σαφής για τη χώρα μας. Και θα με επιτρέψετε πρόεδρε, θα με επιτρέψετε ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές να θυμίσω μια και καλή ότι αυτούς τους έξι μήνες παρουσιάστηκε ουσιαστικά η καθοδήγηση της ε, ε, χώρας μας και θα ήθελα να χαιρετήσω με αφορμή την ομιλία μου εδώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τζόρτζο Ναπολιτάνο, ο οποίος θα αφήσει τα καθήκοντά του μετά από μια μακρά θητεία αλλαγών και έχοντας αντιμετωπίσει αντικσοότητες στην Ιταλία με την ευθεία και την σύνεση που το έχετε αναγνωρίσει και πολλοί από εσάς. Και με πολλές αφορμές αυτήν εδώ την αίθουσα τα περασμένα χρόνια. Στο εξάμεινο αυτό η Ιταλία ε, επεδίωξε δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, να δώσει πολιτική αξία στη δική σας τη δουλειά, κύριε και κύριοι βουλευτές. Στις 2 Ιουλίου, όταν ήρθαμε εδώ για την έναρξη του εξαμήνου, η νέα Επιτροπή δεν είχε ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά της. Εμείς υπήρξαμε πρωταγωνιστές με όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις σε μια επιλογή την οποία θεωρώ ιστορική σημασίας έγινε η επιλογή να δοθεί πολιτική αξία και σημασία στο αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Μαΐου. Ο διορισμός του Ζαν Κλοντ ως Προέδρου της Επιτροπής δεν γεννάται μόνο από την αναγνώριση των αποτελεσμάτων των εκλογών, που από μόνο του θα ήταν ίσως αρκετό διότι σε κάθε περίπτωση ε, ο σχηματισμός που εκπροσώπησε ο κύριος Γιούνκερ δεν μπορούσε να το εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης. Όχι, ήταν μια πολιτική συμφωνία με σίγμα κεφαλαίο που επιβεβαίωσε την επιλογή του κυρίου Γιούνκερ ώστε να δοθεί αξία στην ψήφο των πολιτών, διασυνδέοντας ε, τα καθήκοντα της νέας Επιτροπής Γιούνκερ με ένα, μια δέσμη μεταρρυθμίσεων, με πολιτικά οράματα για τα επόμενα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην ιστορία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεν είναι η πρώτη και α, παρόλα αυτά, μάλλον είναι η πρώτη φορά και θα πρέπει να καταγραφεί στα πολιτικά μας ήθη ε, ακόμη ε, και αν κάποιος το θεωρήσει απλώς ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Η Ιταλία όμως έτσι προτείνει και μια αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο που τα τελευταία χρόνια χαρακτήρισε τις συζητήσεις ε, στην Ευρώπη η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει ρυθμό στα θέματα της ε, ε, οικονομίας. Αλλιώς θα γίνουμε ουραγός σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα. Ε, ήδη ο κύριος Γιούνκερ το συζήτησε αυτό, το έθεσε στα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων και βρίσκω χαρακτηριστικό ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για το πρόγραμμα επενδύσεων και το στρατηγικό πρόγραμμα ευρωπαϊκών επενδύσεων. Δύο προτάσεις για τις οποίες εμείς έχουμε θετική αποτίμηση. Πιστεύουμε ότι στοχεύουν στη σωστή ε, κατεύθυνση. Κατά την άποψή μας πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα και εμείς θα αναλάβουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνη. Είμαστε έτοιμοι να φανούμε γενναιόδοροι με αυτό το ταμείο και να στηρίξουμε τις επενδύσεις για την ε, ευελιξία. Γιατί εάν δεν υπάρξει και ευελιξία, πολλές είναι οι χώρες από τις οποίες προερχόμαστε και προέρχεστε που δεν θα βρίσκονται στις οικονομικές συνθήκες που θέλουμε σήμερα. Η ανοικοδόμηση στη Γερμανία δεν θα ήταν απλή εάν δεν υπήρχε η γενεοδορία όταν έπρεπε, εάν δεν υπήρχε ευελιξία ή πολιτική δεν θα υπήρχε σε αυτήν την αίθουσα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το εξάμεινο αισθανόμαστε ότι υπήρξε βαθιά αλλαγή στην πορεία μας. Δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως να θυμίσω τις συζητήσεις τον ε, Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο με τους ε, εκπροσώπους, φίλους εκπροσώπους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όταν μιλήσαμε για τη σημασία της ανάπτυξης, τη σημασία των επενδύσεων, της αλλαγής όμως της επενδύσεις και τη σχέση των επενδύσεων με την ευελιξία. Μόνο έξι μήνες πέρασαν, αλλά πόσα φαίνεται να έχουν αλλάξει. Αυτά είναι τα δύο αποτελέσματα που νομίζω μπορούμε να τα δούμε ε, από κοινού. Επενδύσεις στην πολιτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιλέγει τη σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε διαμακρών τα αποτελέσματα, ε, το κλίμα, η συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια, η πολιτική της μετάβασης από το Μάρε από την επιχείρηση Μάρε Nostrum στον Τρίτονα, η εξωτερική μας πολιτική σε αντίξωες, αρνητικές ε, συνθήκες, η αυτόματη ε, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η συμφωνία για την συνεργασία μας στην εξωτερική πολιτική, ο αποχαρακτηρισμός που ε, εμπορικών διαπραγματεύσεων, οι γενετικώ τροποποιημένοι οργανισμοί, υπήρξαν και κάποιε κάποια αρνητικά σημεία. Θεωρώ, πρόεδρε Σούλτ, ότι για το Made in η δέσμευση του Κοινοβουλίου αυτού του θεσμικού οργάνου από τον περασμένο Απρίλιο έδωσε τη σωστή όθηση, ζητώντας από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρουν τα απαραίτητα αποτελέσματα. Αυτό δεν έγινε δυστυχώς πραγματικότητα και εκεί είναι ανεξήγητες οι αντιστάσεις κάποιων κρατών μελών. Και να σας, για να καταλάβετε, σας παρουσιάζω αυτό το έγγραφο, έγγραφο που παρουσιάζει τα αποτελέσματα του τελευταίου εξαμήνου εφόσον θέλετε τις λεπτομέρειες και να περάσω τώρα ε, στο δεύτερο μέρος των όσων ήθελα να σας πω. Δηλαδή στο ζήτημα ουσίας. Πετύχαμε αυτούς τους έξι μήνες να δώσουμε πάλι πνοή στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς σε αυτό το ερώτημα. Τη στιγμή που η συζήτηση για το βαθύτερο νόημα της Ευρώπης αντιπαραβάλλεται με έναν άκρατο λαϊκισμό αυτή τη στιγμή αναζητώντας την ελπίδα στην Ευρώπη, όπως με την παρουσία του ο Πάπας Φραγκίσκος φρόντισε να θυμίσει εδώ κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, μιλώντας για την ομορφιά και την ελπίδα που όλοι αναζητούμε. Την Ευρώπη ως κάτι που θα χρησιμεύσει κάτι στον υπόλοιπο κόσμο και καταπολεμώντας τον λαϊκισμό. Την ανάγκη να ε, ριζώσουν οι αξίες μας σε ένα ε, συγκεκριμένο πλαίσιο που όμως δεν θα πρέπει να γίνει απλώς ε, οχυρό. Όχι, θέλουμε να είναι μια αγορά, ένας τόπος συζήτησης η Ευρώπη, όχι ένα οχυρό. Ε, αυτά που εκπροσωπούν την Ευρώπη είναι τα μουσεία και τα σχολεία. Δεν είναι ο φόβο. Η Ευρώπη και η λέξη κλειδί που χαρακτηρίζει την Ευρώπη δεν είναι η ήττα και η σύγκρουση. Είναι ο διάλογο και η συνάντηση. Με αυτή την εφορμή, επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να είμαι πολύ σαφή. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είχαμε κηρύξει την έναρξη, έναρξη του ε, εξαμήνου με την νεαρή εκείνη γυναίκα, την Μίριαμ στο Σουδάν, να είναι κρατούμενη για τις θρησκευτικέ της πεπιθήσεις. Είμαι υπερήφανος που σήμερα η Ευρώπη, κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, επέτρεψε σε αυτή τη γυναίκα να ξαναβρει την ελευθερία της, να πάρει το παιδί της που γεννήθηκε στη φυλακή και να βγει για να ζήσουν μαζί ελεύθεροι, γιατί η Ευρώπη πάνω απ' όλα εκπροσωπεί την ελευθερία. Επιτρέψτε μου, πρόεδρε, να σα πω ότι είμαι συγκινημένος. Συγκινούμε όταν σκέφτομαι ότι στις 20 Αυγούστου και στο δικό σα το όνομα είδα αυτήν την δραματική ιστορία, ε, την όμορφη ιστορία όταν τόσοι ε, νεαροί η ε, στη γενοκτονία της Εμπρένιτσα δεν είχε κάνει τίποτα η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει το τι συνέβη. Δεν είπε τίποτα. Έχει αλλάξει η στάση μας απέναντι στη βία και στις γενοκτονίες. Τώρα έχουμε απέναντί μας τέτοιες περιπτώσεις όπου διαπράττονται περιπτώσεις σοβαρότατων σφαλμάτων και πόνου. Η Ευρώπη εκεί πρέπει να είναι παρούσα. Και πρέπει να θυμηθούμε κυρίες και κύριοι ότι οι πολίτες που κατέβηκαν στους δρόμους του Παρισιού το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Η ιστορική φωτογραφία της Ευρώπης δεν είναι η φωτογραφία των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων που κρατάμε ως ανάμνηση. Όχι. Η φωτογραφία που γράφει ιστορία είναι η φωτογραφία αυτού του λαού, του γαλλικού λαού, που στην ε, ιστορία του με τους καθεδρικούς ναούς, ε, με την ιστορία αυτή που έχει γράψει και μιας και βρίσκομαι στο Στρασβούργο, ε, στη χώρα της Γαλλίας, να αποτίσω φόρο τιμής και στο γαλλικό λαό και σε όλους τους Ιταλούς για τα όσα συνέβησαν Και να θυμίσω ότι αυτό που είναι το βαθύτερο νόημα είναι αυτή η τρομερή εμπειρία που ζήσαμε στο Παρίσι. Με τη Μασαλιώτιδα να τραγουδιέται ενώ βαδίζαμε. Με την εικόνα γυναικών και ανδρών που δεν παρετήθηκαν, δεν συμβιβάζονται με την ιδέα του τρόμου και του φόβου. Με την παρουσία τους στους δρόμους και τις πλατείες του Παρισιού είπαν ότι είναι πιο ε, ισχυροί από τις απειλές η Ευρώπη. Ότι οι τρομοκρατικές απόπειρες δεν μας τρομάζουν. Ότι αν θέλουμε να είμαστε πιστοί στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καθένας, η κάθε μια από εμά έχουμε καθήκον να εντοπίσουμε έναν εχθρό. Ναι, γιατί εχθροί υπήρχουν, υπάρχουν. Ποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάποιος εχθρός. Υπάρχουν εχθροί αλλά αυτοί που λένε ότι η έχθρα θα πρέπει να βασιστεί στη θρησκεία θα έπρεπε να διαβάσουν μια πολύ σημαντική ομιλία. Ομιλία του Αιγυπτίου Προέδρου. Πολλά από τα ραντεβού, ένα από τα πολλά ραντεβού αυτού του εξαμήνου δεν πρόλαβαν να αναφερθώ στις συναντήσεις που είχαμε στο Κάιρο και στη Ρώμη με τους Αιγυπτίους. Μια από τις σημαντικότερες ε, κάμπες ε, για την ε, ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά την 1η Ιανουαρίου σε ένα πανεπιστήμιο του Καΐρου είπε ότι εχθρός δεν είναι η θρησκεία. Εχθρός είναι εκείνη που κατηγορούν και επιδεικνύουν ως υπευθύνους όσους έχουν θρησκευτικές πεπιθήσεις. Θέλουν να θανατώσουν όμως τη θρησκεία. Είναι η θρησκεία και ο φανατισμός, ο θρησκευτικός φανατισμός λοιπόν. Ο στόχος μας δεν είναι να εθελοτυφλούμε και να μην δούμε τον εχθρό, αλλά να σκεφτούμε ότι να, να αφήσουμε να σκεφτεί κανείς ότι θα μας παραλύσει ο φόβος, ότι μπορεί να μας επιτρέψει να μην δράσουμε. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εγκλωβιστούμε, να δημιουργήσουμε γύρω μας τάφρους προστασίας και να υψώσουμε τύχη. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα φτιάξουμε έτσι την Ευρώπη. Δεν θέλουμε να ζήσουμε φοβισμένοι και, και κρυμμένοι λόγω του φόβου. Όχι. η λέξη ταυτότητα δεν αντίκειται με τη λέξη, δεν αντιφάσκει με τη λέξη ενσωμάτωση. Ως Ιταλός, ως αριστερός, πρέπει να πω ότι δεν θα αφήσουμε την λέξη ταυτότητα στα στόματα όσων φωνάζουν πιο δυνατά. απλώς. όχι, ταυτότητα είναι μια ωραία λέξη που ανήκει σε όλους μας, που εκφράζει το βαθύτερο νόημα της ευρωπαϊκής ύπαρξης. Εγώ είμαι περήφανο για τις ρίζε μου. Είμαι περήφανο για τους δρόμους που έπαιξα ποδόσφαιρο, για τα σχολεία στα οποία φίτησα ως παιδί. Είμαι περήφανο που είμαι Ιταλός, που είμαι Ευρωπαίο, που είμαι από τη Φλωρεντία. Είμαι περήφανο για τα προσωπικά μου βιώματα, γιατί η ταυτότητά μου είναι ένα βαθύ χαρακτηριστικό. Το αντίθετο τη ταυτότητα δεν είναι η ενσωμάτωση. Το αντίθετο τη ταυτότητα είναι η ανωνυμία. Το αντίθετο της ενσωμάτωσης και της ένταξης είναι η κατάρρευση, είναι η καταστροφή, είναι η φθορά. Σήμερα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δύναμη να πούμε με αποφασιστικότητα και πυγμή ότι όταν εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εκτός. Σκεφτόμαστε ότι η υπεράσπιση της ταυτότητάς μας είναι το να εγκλωβιστούμε σε οχυρά και φρούρια στο όνομα της ασφάλειας, ουσιαστικά μειώνουμε τους εαυτούς μας και δεν καταλαβαίνουμε ότι η ελευθερία και η ευθύνη είναι προϋποθέσεις της ασφάλειας. Δεν υπάρχει δυνατότητα ασφάλειας χωρίς ελευθερία. Σε αυτόν τον κόσμο, εχθροί μας, είναι αυτοί που προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο ζωή μα, όχι αυτοί που προσπαθούν να μα σκοτώσουν. Δεν θα το επιτρέψουμε σε κανέναν όμω. Σε κανέναν δεν θα επιτρέψουμε να αλλάξει τον τρόπο ζωή μα. Μπορείτε να το χαρακτηρίσετε με όποιον όρο σα βολεύει αυτό. Πόλεμο, σύγκρουση, όπω σα βολεύει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ε, η εξή το φάσμα της δημαγωγίας μπορεί να φέρει κάποια ποσοστά περισσότερο στις εκλογές, ίσως. Αλλά αν ε, θέλουμε να είμαστε ηθήνουσα τάξη, η πολιτικοί ηθήνοντες, γυναίκες και άντρε, που θα φέρει την Ευρώπη να αλλάξει την πορεία της, να αναλάβει τα καθήκοντά της, για να γίνει αυτή η σοβαρή αλλαγή, η καμπή, πρέπει να πούμε το εξή απλό. Και θα πω το εξή απλό για να κλείσω. Εάν βλέπουμε να αλλάζει τάση η πολιτική σήμερα στην Ευρώπη, αυτό συμβαίνει γιατί αυτούς τους μήνες και αυτά τα χρόνια είδαμε ότι ο κόσμος ζητά περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη, αλλά πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αυτό το είδος Ευρώπης που οικοδομήσαμε αυτά τα χρόνια έχει δώσει την εντύπωση συχνά ότι είναι ένα μοντέλο βασισμένο στην οικονομία, στις παραμέτρους, τους κανόνες και την λιτότητα. Πρόεδρε, στο τέλος αυτών των έξι μηνών νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ήταν λανθασμένη αυτή η στάση. Η αλλαγή που φέρνει η Επιτροπή Γιούνκερ μετά από το εξάμηνο αυτό είναι μια αλλαγή που θα έπρεπε να την έχουμε φανταστεί από έξι χρόνια τώρα, όχι έξι μήνες. Αλλάζει σήμερα ο κόσμος. Προσπαθεί να επενδύσει στο μέλλον. Η Ευρώπη όχι ακόμα. Εμείς πήγαμε στο Brisbane, ε, στο G20 ε, ως Ευρωπαίοι και οι λέξεις καινοτομία και ανάπτυξη ηχούν παντού στον κόσμο. Θέλουμε λοιπόν να αναλάβουμε τα ενία αυτής της αλλαγής και όχι να βρεθούμε ουραγοί. Εάν η Ευρώπη λοιπόν κοιτάξει τον εαυτό της στα μάτια με την επίγνωση ότι είναι υπερδύναμη, όχι οικονομική, αλλά υπερδύναμη αξιών. Την ίδια υπερδύναμη αξιών που κάποιοι από τους λαϊκιστές θέλουν να ακυρώσουν. Και θα ε, αφήσω πια ε, το λόγο στην Λετωνική Προεδρία και τις ευθύνες στη Λετωνική Προεδρία θυμίζοντας ότι το 1955 η Ιταλική Προεδρία ήταν εκείνη που σφράγγισε τη συμφωνία για την άμεση εκλογή του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή αυτή. Πριν από 40 χρόνια η Λετωνία δεν ήταν καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βρισκόταν σε μια τελείως διαφορετική φάση της ιστορίας της. Σήμερα έχουμε δείξει ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να αλλάξει. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η αλλαγή αυτή πρέπει να μας κάνει να στραφούμε και στην πολιτική γειτονία με διαφορετικό τρόπο. Και αυτήν την σφαγίδα θέλουμε να αφήσουμε. Και αυτό το μήνυμα προς τη νέα ε, Προεδρία. Πολιτική γειτονία και προσοχή προς τη Μεσόγειο πρέπει να προσέξουμε την ε, εξωτερική μας πολιτική και με χώρες όπως η Αλβανία, η Σερβία, τη συνεργασία τη χρειαζόμαστε. Δεν μπορεί η συζήτηση ε, περί διεύρυνσης να βασιστεί μόνο στον φόβο. Θα πρέπει να θυμηθούμε τις σχέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας και τις δικές μας μαζί τους. Είναι ένα από τα ευαισθητότερα θέματα αυτού του εξαμήνου και θα χαρακτηρίσει την περίοδο που ζούμε. στις επόμενες λοιπόν διεθνείς ευθύνε της Ιταλία, ξεκινώντας με τη διεθνή έκθεση που από το Μάιο θα καλύψει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στον πλανήτη μας πώς θα αλλάξει η ζωή των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει μια επένδυση στον τρόπο διαβίωσής μας. Αλλά γι' αυτό σας θύμισα από την αρχή τον ε, τηλέμαχο. Ε, βέβαια θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα βιβλία. Για κάποιους από εσά είναι πιο δύσκολο να διαβάσουν πάνω από δύο φαντάζομαι. Αλλά σήμερα πρόεδρε μπορώ να σας πω ότι έμαθα τι σημαίνει η Ευρώπη μελετώντας την ιστορία της πόλης μου. Στην ιστορία της πόλης μου υπάρχει ένα μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, ο Δάντη, ο οποίος όταν επιτρέπει, όταν βάζει τον Οδυσσέα να μιλήσει, ε, του, ε, τον κάνει να λέει λόγια που τα βρίσκω σήμερα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι ιτημένος ο Οδυσσέας, αλλά ο Δάντης, ο Οδυσσέας με το στόμα ε, μέσα από το Δάντη λέει ότι δεν είστε φτιαγμένοι για να ζήσετε στην άγνοια, αλλά για να ζητήσετε την αρετή και την σοφία. Αυτό νομίζω είναι το βασικό μήνυμα για μας σήμερα. Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να επιλέξει εάν θα θελήσουμε να ζήσουμε στην αγνιά μας επιλέγοντας τα μηνύματα και τις ειρήνες του λαϊκισμού που μπορεί κάποια ε, δεκαδικά ψηφία στις εκλογές να τα προσφέρουν αλλά αν θέλουμε να επιδιώξουμε την αρετή και τη σοφία, να είμαστε Ευρωπαίοι και να κινούμαστε βάσει της καρδιάς μας και των ευθυνών μας, τότε θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ευρώπη είναι η αρένα για τις προκλήσεις του αύριο. Θα ήθελα με αυτό να ευχαριστήσω λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο και να πω και πάλι ότι η Ιταλία πιστεί στο μήνυμα του πολιτισμού, των αξιών και των ιδανικών θα συνεχίσει να εργάζεται για μια Ιταλία των λαών και μια ε, Ευρώπη που θα είναι λιγότερο η Ευρώπη της γραφειοκρατίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Κόμπερν, 12 φορές ξεστομίσατε τον όρο rubbish, ideas. Θα αρχίσει να πιστεύει ο κόσμος ότι αυτό είναι το όνομά σας. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιούνκερ. Sehr verehrter Herr. κύριε Πρόεδρε. Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, από καιρού εις καιρών υπάρχουν στιγμές που είναι πραγματικά δύσκολο να περάσει κανείς από τη μία φάση στην άλλη. Εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε σήμερα στην ε, ελευθέρωση των ε, νεζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αυτοί που γεννήθηκαν πολύ μετά τον πόλεμο και αυτοί που γνωρίζουν τα γεγονότα στα οποία αναφερθήκατε μόνο από τα βιβλία δεν μπορούν να αντιληφθούν τον πόνο που μάστησε την Ευρώπη όχι μόνο την περίοδο 40 με 45 αλλά 33 με 45 θα έλεγα. Προσοχή λοιπόν στη λάθος εκκίνηση. Να μάθουμε από την ιστορία μας, να πάρουμε τα μαθήματα που πρέπει από αυτήν. Σήμερα λοιπόν Βρισκόμαστε εδώ, στη γαλλική επικράτεια. Πώς να ξεχάσει κανείς αυτές τις στιγμές το δράμα, την τραγωδία, τη συλλογική και ατομική τραγωδία που έζησε η Γαλλία στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε σοκ, να, ιδιάζουμε, να γανακτούμε από τα όσα έλαβαν χώρα στο Παρίσι αυτή τη βδομάδα. Είμαστε όλοι σαρλί, αλλά μέσα στον κόσμο υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, πολύ σαρλί. Είμαστε όμως στη Γαλλία και επειδή βρισκόμαστε στη Γαλλία θα πω ζήτω η δημοκρατία και ζήτω η Γαλλία. Έχουμε φτάσει στο τέλος της Ιταλικής Προεδρίας και τις παραμονές της Λετωνικής Προεδρίας. Είναι μια στιγμή η οποία μας καλεί να προβληματιστούμε και να πάμε ακόμα πιο πέρα. Αυτή είναι η όρη της Ιταλικής Προεδρίας, μιας χώρας ιδρυτικού μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αύριο θα ακούσουμε την Λετωνό Πρωθυπουργό. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί το 1957 ότι το 2015 η Λετωνία θα προείδρευε τον... την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήταν επικεφαλής του προορισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο συμβολίζει τη συμφιλίωση της, ε, στα πλαίσια της ιστορίας και της γεωγραφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καθορίσει το τέλος εκείνου του δόγματος της ε, Ευρώπης πριν από πολλά χρόνια που ήταν κατά της εφηλίωσης αυτής. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα λέω ζήτω η Ευρώπη γιατί αύριο όπως και σήμερα ζούμε μια πολύ μεγάλη στιγμή στην ευρωπαϊκή ιστορία και μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όσα κάναμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της Ιταλικής Προεδρίας, την οποία, την οποία θέλω να ευχαριστήσω. Αγαπητέ φίλε, θέλω να σε ευχαριστήσω και να σε συγχαρώ. Κατά τη διάρκεια της υπουργικής μου ζωής, πέντε φορές ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου. Γνωρίζω το αίσθημα αυτό όταν φτάνει κανείς στο τέλος της προεδρίας του, του εξαμήνου του. Νιώθει ανακούφιση, νιώθει ικανοποίηση που μπορεί να δώσει στη σκητάλη στην επόμενη προεδρία. Από την άλλη μεριά όμως νιώθουμε και μια κάποια απογοήτευση γιατί δεν καταφέραμε να κάνουμε όλα όσα ονειρευτήκαμε στην αρχή της προεδρίας μας. Έτσι λοιπόν και η Ιταλική κυβέρνηση έκανε πολλά πράγματα πολλά τα οποία μας βοήθησαν να συμφωνήσουμε. Για παράδειγμα για τον προπολογισμό ε, του 2015. Και από αυτού η συνεργασία και η συνενοχή κατά κάποιο τρόπο ε, μεταξύ μας μας βοήθησε όλους μαζί να συμφωνήσουμε με το άλλο σκέλος ε, του προϋπολογισμού, το Συμβούλιο για τον προπολογισμό του 2015. Αν δεν είχαμε την καθημερινή βούληση της Ιταλικής Προεδρίας, το αποτέλεσμα αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Αν η Ιταλική Προεδρία δεν έκανε όσα κατάφερε να κάνει, σήμερα δεν θα βρισκόμασταν στη θέση που βρισκόμασταν, αλλά θα ήμασταν μέσα σε μια δημοσιονομική κρίση με τις επιπτώσεις βέβαια που γνωρίζουμε. Η Ιταλική Προεδρία λοιπόν κατάφερε και βοήθησε να εγκρίνουμε όλες τις νομικές πράξεις που έπρεπε να έχουμε εγκρίνει και για τον ε, μηχανισμό εξυγίασης που αποτελεί πλέον τη βάση της Τραπεζικής Ένωσης. Και καταφέραμε ως ε, Προεδρία βέβαια να στηριχτούμε και στην ε, βούληση της Ιταλικής Προεδρίας που ήταν να προχωρήσουμε γρήγορα και στις επενδύσεις. Κατά την προεκλογική εκστρατεία και όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπαμε ότι θέλαμε δημοσιονομική παγίωση, μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές που είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά θέλουμε και μία διάσταση ανάπτυξης και απασχόλησης. Αυτό είναι το τρίγωνο αρετής που θέλαμε να εφαρμόσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή Τη οποία είμαι επικεφαλή. Χωρί λοιπόν την ενθάρρυνση από πλευρά ε, τη Ιταλική Προεδρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω να μην τα είχε καταφέρει να προχωρήσει τόσο γρήγορα όπω τα κατάφερε για να βάλει και πάλι την ανάπτυξη στην πρώτη γραμμή που αποτελεί μια βασική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών και ολόκληρη τη Ευρώπη. Το είπε και ο Ματέο, σήμερα το απόγευμα το Σώμα των Επιτρόπων θα επανέλθει στα νομικά κείμενα προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το επενδυτικό ταμείο. Και σήμερα θα έχουμε και ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και για αυτό το σημείο, αλλά και για άλλα, προχωράμε χάρη στον ενθουσιασμό της Ιταλικής Προεδρίας. Μας έχει εμπνεύσει πολύ εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δράση της Ιταλικής Προεδρίας. Για να γίνω πιο κατανοητός, θέλω να πω πως ναι, η Ιταλική Προεδρία έκανε καλή δουλειά, μπομπούλο όπως λέμε στα γαλλικά, και η Ιταλική κυβέρνηση όταν θα έχει φύγει από την Προεδρία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα συνεχίσει να εμπνέεται από τόσα έκανε κατά τη διάρκεια του Ιταλικού εξαμήνου και θα παραμείνουμε όλοι σε αυτό το πνεύμα. Βίβα Ιταλία! Ζήτω Ιταλία! Σας ευχαριστώ. Κύριε Γιόνκερ και τώρα εκ μέρους Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο συνεχίζουμε τη συζήτηση. Θα ακούσουμε τον κύριο Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή, απερχόμενε Πρόεδρε τη Ιταλική Προεδρία. Κυρίε και κύριοι, έχει μεγάλη σημασία στην Ιταλία, η Ιταλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο εμπορικά, βιομηχανικά, πολιτιστικά. Είναι ένα κομμάτι του κοινού ευρωπαϊκού μα οίκου. Και γι' αυτό είχαμε πολλέ προσδοκίε για την ε, Ιταλική Προεδρία. Ήταν υψηλέ οι προσδοκίε όταν ξεκινούσε πριν από ένα εξάμηνο η Ιταλική Προεδρία. Και πρέπει να πω, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, για τα αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να διαπιστώσουμε τώρα με μια σταθερή δημοσιονομική πορεία, ότι τα οφείλουμε και στην προσπάθεια τη Ιταλική Προεδρία. Σταθερότητα και ισχύ. Έθεσε το θέμα τη μετανάστευση η Ιταλική Προεδρία ο Υπουργό των Εσωτερικών Αντζελίνο Αλφάν, ήταν εκείνο ο οποίο έφερε στο θεματολόγιο και την ημέρη διάταξη το θέμα αυτό που ε, υποχρεώνει τους Ευρωπαίους να αντιληφθούν ότι πρόκειται για μια κοινή υποχρέωση και τα θέματα των σχετικών επενδύσεων. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά για τη συνεργασία, για τη δουλειά σας, για την συμμετοχή όλων των Υπουργών και των τεχνοκρατών σας. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην ιστορική και δημοκρατική διάσταση της τελευταίας ε, περίοδου το ότι θέσατε εσείς δηλαδή ε, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το ερώτημα ποιος ηγείται της Ευρώπης. Το οφείλουμε σε εσά το γεγονός ότι ο ψηφοφόρος είναι αυτός ο οποίος εκλέγει και τον πρόεδρο της Επιτροπής ακόμη. Το γεγονός ότι σήμερα κάθεται εδώ ο Ζων Κλοντ Γιούνκερ εκλεγμένος άμεσα από την ψήφο του Ευρωπαίου πολίτη το οφείλουμε σε έναν βαθμό και σε εσά. Κλείνει λοιπόν το εξάμεινο τώρα της Ιταλικής Προεδρίας. Μιλήσαμε για, το εξάμεινο, για την ε, ε, διελκυστίνδα ευελιξία, ανάπτυξη, λιτότητα. Είπατε ότι πρέπει να κοιτάμε όχι μόνο τους οικονομικούς όρους αλλά και τις αξίες. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Γιατί πρέπει να στηριζόμαστε πάντα σε μια διελκυστίνδα, σε μια σύγκρουση. Γιατί να μην κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούν και με βάση τις αξίες βεβαίως να ενισχυθούν οι προσπάθειές μας και να οικοδομήσουν κάτι καλύτερο με τις αξίες της Ευρώπης να ενισχύσουμε την οικονομία, την οικονομία μας. Όχι λοιπόν διαπάλι, όχι λοιπόν διαλκυστίνδα, αλλά να υπογραμμίσουμε αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Και όταν ε, παρουσίασε ο Jean-Claude Juncker ε, την πρότασή του για το, για το πακέτο των επενδύσεων και θα το εξηγήσει σήμερα το απόγευμα στις νομοθετικές του διαστάσεις είπατε ότι πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο σημαίνει επενδύσεις, ναι βεβαίως, και ανάπτυξη, ναι βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα και μεταρρυθμίσεις για τη σταθεροποίηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες δημοσιονομικές. Και όταν γίνει η πρόταση σήμερα θέλουμε να ακούσουμε πιο συγκεκριμένα τι θα σήμαινε όρος ευελιξία. Είπατε και εσείς κύριε Ρέντσι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι οι κανόνες, το six-pack, το two-pack, τα, δύο τα σύνολα των έξι και των δύο νομοθετημάτων δεν πρέπει να διαταραχθούν, θα πρέπει να ισχύσουν ως έχουν. Αυτό μαζί με την ευελιξία είναι μια πολύ σημαντική πρόταση και πρέπει να το δούμε έτσι. Έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει σήμερα το απόγευμα τι σημαίνει ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα και αυτό που αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι οι κανόνε δεν αλλάζουν. Πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα στην Ευρώπη και για να αποδείξουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι ω Ευρώπη και στον άνθρωπο και στον πολίτη και στον εξωκόσμο. Επίσης η σημερινή εβδομάδα κύριε και κύριοι έχει μια διαφορετική γεύση θα έλεγα γιατί είμαστε όλοι πολύ βαθιά επηρεασμένοι από τα γεγονότα του Παρισιού και τις επάνθρωπες επιθέσεις. Νομίζω ότι οφείλω τώρα να κλείσω υπογραμμίζοντας αυτό το οποίο μας ενώνει όλους τους Ευρωπαίους. Τις αξίες του ανθρώπου. Αυτά τα διαπραγμάτευτα της Ευρώπης μας, της Υπήρου μας, της Δύσης. Ότι Δύση δεν είναι οι ακραίες θέσεις ορισμένων. Δύση είναι ένωση, επικουρικότητα, διαφωτισμός, αποδοχή, διαλλακτικότητα. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη Δύση, το δυτικό πολιτισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πιτέλα εκ μέσω Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κύριε Πρόεδρε Ρέντσι, στις 2 Ιουλίου του 2014, στην έναρξη της Ιταλικής Προεδρίας και στην παρουσία σας εδώ, είχατε πει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξαναβρούμε την πνοή, την ψυχή της Ευρώπης. Την Κυριακή πήγαμε στο Παρίσι η ψυχή της Ευρώπης ήταν εκεί. Εκατομμύρια άνθρωποι. Για αυτούς που θέλουν να μας κλείσουν στα σπίτια μας και να υψώσουν τύχη, να εμπνεύσουν τον φόβο και την καχυποψία, την Κυριακή απαντήσαμε. Απαντήσαμε βγαίνοντας τους δρόμους, βαδίζοντας ενωμένοι οι επιθέσεις στο Παρίσι δεν ήταν απλώς επιθέσεις κατά της ελευθερίας, της σκέψης και της έκφρασης. Ήταν επίθεση κατά της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Και ευρωπαϊκή κυριαρχία σημαίνει ότι ένας λαός είναι ελεύθερος να επιλέξει πώς θα ζει και κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει σε εμά τουλάχιστον το πώς θα ζούμε. Προσοχή λοιπόν να μην πέσουμε στην παγίδα της τρομοκρατίας. Την τρομοκρατία που θέλει να μετατρέψει τις κοινωνίες μας σε φρούρια που να βρίσκονται σε πολιορκία μετά τις 11, την 11η Σεπτεμβρίου, η Αμερική αποφάσισε να χτίσει περισσότερες φυλακές παρά κολέγια. Μην κάνουμε το ίδιο σφάλμα εδώ στην Ευρώπη η Ευρώπη θέλουν να ζουν σε μια κοινωνία ανοιχτή, όπου η ελευθερία και η ασφάλεια να βαδίζουν χέρι-χέρι. Για να ξαναβρούμε την ψυχή της Ευρώπης, δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στα λόγια και τις ρητορίες. Πρέπει να ασχοληθούμε με τις πραγματικές ζωές των ανθρώπων, με τα άγχη και τις ε, ελπίδες τους. Δηλαδή, να δώσουμε στους πολίτες μια ζωή ελεύθερη και με αξιοπρέπεια. Η πρώτη ελευθερία είναι να καλύψουμε τις ανάγκες. Η και κοφεύουσα ε, λιτότητα που δίνει έμφαση στην επισφάλεια και την φτώχεια είναι αυτό που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Η Ιταλική Προεδρία λοιπόν έδωσε στην Ευρώπη τα όπλα για να ξαναπεράσει στη σωστή πορεία. Όταν τον Ιούλιο μιλήσαμε για επενδύσεις που θα πρέπει να ανακάμψουν, πολλοί είχαν χαμογελάσει τότε κύριε Πρόεδρε. Αλλά ε, πολύ, ε, σήμερα το απόγευμα κιόλας, όπως θυμήσατε και εσείς ο ίδιος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει για συγκεκριμένο κανονισμό για το πρόγραμμα των 300 δις. Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και με πολλά ισχυρά σημεία και με κάποιες αδυναμίες. Η δική μας η ομάδα ούτως ή άλλως έχει αναλάβει δέσμευση να ε, παρέμβει για να τροποποιηθούν αυτά. Και σε αυτό το εξάμεινο ανασκόπηση μιλήσατε για την ευελιξία που επιδιώξατε. Τι είναι αυτή η ευελιξία που επιδιώκει ο Ρέντσι, είπανε πολύ ηρωνικά. Φαινόταν σαν μια, σαν μια μάχη του Δον Κιχώτη, με, τους, ε, με τον Δον Κιχώτη που δεν ξέρουμε εάν θα καταφέρει να εξαρθρώσει αυτή την λιτότητα που είναι η βάση του συμφώνου. Όχι, η Επιτροπή σήμερα παρουσιάζει συγκεκριμένε προτάσει για την ευελιξία και πιστεύω ότι θα συμπεριλαμβάνονται σημαντικά στοιχεία για τα οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Χάρη και στην Ιταλική Προεδρία πετύχαμε να ανακόψουμε ε, όσου ήθελαν ε, τα κράτη-μέλη να γίνουν υπόλογα μόνο με πρόστιμα και με κυρώσεις γιατί δεν ε, εφάρμοσαν πλήρως τα όσα επέβαλαν οι Βρυξέλλες. Όχι. Αυτό έγινε ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρία και θεωρούμε πολύ σημαντικό. Ο χρυσό κανόνα των επενδύσεων έμοιαζε όνειρο, σήμερα. Όχι. Ο χρυσό κανόνα είναι μια μάχη ιστορική που κέρδισε η ομάδα μα. Η συγχρηματοδότηση των επενδύσεων στην Ευρώπη. Οι επενδύσει που προβλέπει το πρόγραμμα ε, του κ. Κιούνκερ ε, δεν θα ανακοπούν από το σύμφωνο τη σταθερότητα για όσου δεν βρεθούν πάνω από το όριο του 3% του ελλείμματο. Και η συγχρηματοδότηση των διευθυντικών ταμείων. Και αυτό έφταζε, έμοιαζε όνειρο, χήμερα. Όχι, τώρα έγινε γεγονό. Είναι ένα επαναστατικό στοιχείο. Ναι, πηγαίνετε. Πηγαίνετε να τα πείτε στου πολίτες με τους ε, τοπικούς φορείς, με τις ε, περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ναι, θέλουμε περισσότερα βεβαίως αλλά αυτά είναι ήδη γεγονότα που έχουμε αποσπάσει. Είναι συγκεκριμένα στοιχεία. Επιτρέψτε μου ένα παράθεμα, ε, ε, κύριε Σούλτ. Σε ένα αφήγημα, του λέει, ε, λέει ένα παιδί σε ένα γέροντα αν μπορεί να αγγίξει τα, στάρια, τα αστέρια. Και του λέει ο γέροντας ότι μόνο εφόσον τα πόδια του πατάνε στέρεα στη γη μπορεί να αγγίξει τα αστέρια. Έτσι με τη δική σας Προεδρία, με εσά κύριε Ρέντσι, καταφέραμε να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να πάρει μια τροπή και ένα όραμα για το μέλλον. E Εκ μέρου τη Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μισθών, ο κύριο Λεγκούτκο. Uh, e Κύριε Πρωθυπουργέ Ρέντζο, αναρωτηθήκατε στην αρχή της Προεδρίας σας πώς θα μοιάζαμε αν παίρναμε σέλφι τους αυτούς μας. Εγώ αναρωτιέμαι ο Ιταλός Πρωθυπουργός πώς θα μοιάζε σήμερα να έπαιρνε ένα σέλφι. Έβγαζε μια τέτοια φωτογραφία τον εαυτό του θα έλεγα ότι δεν θα υπήρχε και πολύ περιεχόμενο. Και δεν εκπλήσει, γιατί από την αρχή θα επρόκειτο για μια πολύ μινιμαλιστική ατζέντα όσον αφορά την κατάσταση μετά τις εκλογές. Πώς κατάφερε λοιπόν να πετύχει συμφωνίες στη, στο νομοθετικό τομέα η Ιταλική Προεδρία με το Συμβούλιο, πρώτα απ' όλα για την νομοποίηση του παράνομου χρήματος. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι η συμφωνία με τη σχετική οδηγία βάζει δυσκολίες και στους απλούς ανθρώπους οι οποίοι μπλέκονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας αλλά από την άλλη μεριά τις εκατομμύρια ευρώ καταλήγουν σε εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις. Δεύτερον, ε, γενετικά τροποποιημένα ε, προϊόντα, οργανισμοί. Και αυτό είναι ένα θέμα που διχάζει πολύ και δείχνει ότι κάποιες κυβερνήσεις είναι υπέρ αυτών και άλλες δεν είναι. Τρίτον, προπολογισμό 2015. Πράγματι, συμφωνήθηκε ο προπολογισμό αυτό, αλλά νομίζω ότι εξακολουθούν να μένουν πολύ απλήρωτοι λογαριασμοί. Και εδώ χάθηκε η ευκαιρία να δώσουμε μια υπεύθυνη απάντηση και αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. Έπειτα μετανάστευση στη Μεσόγειο, αυτό εσείς το θεωρείτε θετικό. Πέμπτον, οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, το Και εδώ δεν ξέρουμε πολλά για τις οδηγίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Για να ξέρουμε κατά πόσο μπορούν να καθισχαστούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι βαθμό θα σας έβαζα. Θα σας έβαζα καλός. Δεν θα σας έβαζα άριστα. Συγχαρητήρια παρόλα αυτά. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των φιλελευθέρων, ο πρόεδρος κ. Φερχόφστατ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρέντσι, καταρχάς είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την φιλοευρωπαϊκή σας τοποθέτηση. Για να είμαι ειλικρινής, ανησυχώ κάπως με την Ιταλία. Όταν βλέπω από τις δημοσκοπήσεις τα τρία κόμματα, τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης που συγκεντρώνουν ένα 40 περίπου 100 όπως είναι φυσιολογικό στη δημοκρατία είναι κόμματα που στρέφονται κατά του ευρώ και της ε, ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό εύχομαι να επιτύχετε στις μεταρρυθμίσεις σας στην Ιταλία ώστε να σταματήσετε αυτά τα αντιευρωπαϊκά κινήματα στη χώρα σας γιατί τη χρειαζόμαστε την Ιταλία, πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ευχαριστώ και τον κύριο Γκότσι για την πολύ συγκεκριμένη δουλειά Επίσης θέλω να τιμήσω τον Τζόρζο Ναπολιτάνο για την ε, μεγάλη του συμβολή. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσετε και εσείς για το Κοινοβούλιο που έδωσε το, ε, την κατεύθυνση της Προεδρίας. Νομίζω, όπως είπε και ο κύριος Βέμπερ, έχουμε πλέον ε, φτάσει στο τέλος αυτής της συζήτησης για το αν πρέπει να έχουμε την ε, πειθαρχία ή την ευελιξία. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται και τα δύο και αυτό ε, σημαίνει βέβαια τέλος της συζήτηση, αλλά ταυτόχρονα αρχή της δουλειάς που πρέπει να γίνει γιατί χρειάζεται αυτό το σχέδιο επενδύσεων. Και πρέπει να σας πω κύριε Ρέντσι ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα και ελπίζω ότι θα έχω στο προσεχές συμβούλιο και τη δική σας υποστήριξη είναι ότι δεν μπορούν όλοι να μπουν υπό κάθε όρον στο, σχέδιο επενδύσεων αυτού του επενδυτικού σχεδίου. Δεν μπορεί αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος στα κράτη-μέλη να μην μπουν στο σχέδιο των επενδύσεων για να στηρίξουν το επενδυτικό αυτό σχέδιο και να, το να εξασφαλίσουν την επιτυχία του. Είναι απαράδεκτο το να λένε κάποια κράτη-μέλη όχι, όχι, εμείς δεν εμπλεκόμαστε, δεν είναι δική μας δουλειά. Επίσης χρειαζόμαστε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όχι απλώς την ανακοίνωση των μεταρρυθμίσεων, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και χρειαζόμαστε ένα πακέτο νομοθετικό για να ανοίξουν αυτές οι κύριες αγορές, αλλά είναι κάτι που θα συστήσουμε αργότερα με την Επιτροπή. Ένα πράγμα όμως με απογοητεύει και πρέπει να το πω στην Ιταλική Προεδρία, για να είμαστε και ειλικρινείς μέσα, είναι το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες, το ότι δεν ολοκληρώθηκε το πακέτο αυτό. Α είμαστε ειλικρινεί. όλοι μιλούμε για επενδύσεις, ψηφιακό κόσμο, Google και απάντηση στην Google και όλα αυτά. Ε, σήμερα, 2015, δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε με τα κράτη-μέλη για την ψηφιακή αγορά και το πακέτο για τις ε, τηλεπικοινωνίες. Να σταματήσουν οι επιβαρύνσεις για το roaming, να υπάρχει μια μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτών. Ε, αυτή είναι η απογοητευσή μου. Ελπίζω όμω και με την πίεση βέβαια και των Ιταλών η επόμενη Προεδρία και το επόμενο εξάμεινο να φέρει πραγματικέ αλλαγέ στην ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ. εκ μέρους τη ομάδα, της Νοτική αριστερά, Ο κύριος Μαλτέζα έχει το λόγο. Πρόεδρε, εκεί στο Παρίσι εκατομμύρια πολίτες έκαναν να χτυπήσει η καρδιά της Ευρώπης. Και είδαμε δίπλα-δίπλα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να βρίσκονται μαζί στι ίδιε πλατείε. Πριν από 6 μήνες όμως μας είχατε πει ότι έχετε τη μαγική συνταγή για να φέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες πιο κοντά σε ένα θεσμικό όργανο που χαρακτηρίσει ανιαρό εσείς. Ενεργεία, τόλμη και θάρρος χρειάστηκαν, το αναγνωρίζω, αλλά όλα αυτά παρέμειναν κενά λόγια τους τελευταίους αυτούς έξι μήνες αναζητήσατε μικρές ε, οδούς διαφυγής με τέτοιες συμφωνίες που στις λεπτομέρειές τους θα μπορούσαν να δώσουν την αυταπάτη. Αλλά αυταπάτη γιατί, ότι η Ιταλία με το τρίτο κρατικό χρέος στον κόσμο θα μπορέσει να ξεφύγει με μερικούς κανόνες ευελιξίας από το σύμφωνο σταθερότητας. Η Ιταλική πραγματικότητα διαφέρει από το πεπρωμένο μιας περιφέρειας μιας μεγάλης αυτοκρατορίας δεν είχατε την τόλμη να ζητήσετε το, τον τερματισμό της λιτότητας. Ε, το εξάμεινο αυτό ήταν πολύ λιγότερο ευρωπαϊκό παρά ιταλικό. Εσείς ασχοληθήκατε με το να δείχνετε αγωγές ομοιοπαθητικής ε, στους Ιταλούς όπως ε, την καταπολέμηση της ενεργείας με μαζικές απολύσεις ή την έγκριση δημοσιονομικών συμφώνων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πριν από έξι μήνες ο κ. Φερχόφστατ είχε πει ότι στη σχέση Ιταλίας-Ευρώπης είχαν χαθεί τουλάχιστον 10 χρόνια με τις ανοησίες του Μπερλουσκόνη. Τώρα έχουμε φτάσει τα 10 χρόνια συν 6 μήνες. Εκ μέρους των Πρασίνων η Πρόεδρος κυρία Χάρμς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. κύριε, Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ Ρέντσι, ξέρω ότι η Προεδρία σας δεν ήταν απλή υπόθεση. Είχατε στα χέρια σας την Προεδρία στη φάση αυτή της μετάβασης. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε λοιπόν πάρα πολλά. Θα ήθελα να ήσασταν πολύ πιο ανοιχτοί ε, στην συζήτηση των προβλημάτων που εκδηλώθηκαν ή ξανέρθαν στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι εχθές συζητήσαμε ξεκάθαρα και είπαμε ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους πολίτες της Γαλλίας γιατί με αυτή τη Μάρσχα Επιπλικέν, με την πορεία για τη δημοκρατία έδωσαν μια νέα ευκαιρία στον κόσμο να ξαναδεί και να ξαναορίσει τις αξίες, τους στόχους, τις σχέσεις πολιτείας και πολίτη. Όλα αυτά που συζητούμε εδώ και καιρό. Και εάν προσμετρήσουμε την επιτυχία σας με βάση τους στόχους της Προεδρίας σας, πρέπει να ξανασυζητήσουμε τώρα πώς η δυσπιστία θα γίνει εμπιστοσύνη. Και αυτό όχι μόνο μεταξύ διαφόρων ομάδων πολιτών της κοινωνίας μας, αλλά πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των πολιτών προς την πολιτεία. Και ε, είπατε πώς ε, βλέπετε την απάντηση που θα πρέπει να δώσουν οι Υπουργοί των Εσωτερικών ε, στην, στο θέμα της ελευθερίας στην Ευρώπη. Είδα εγώ πόσα ήταν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές για τους δολοφόνους αυτούς που έκαναν τις επιθέσεις. Πόσα, πόσα, πόσα στοιχεία. Και τώρα με ανησυχία διαπιστώνω ότι ζητάτε ακόμα περισσότερα στοιχεία παρότι δεν είχαν μπορέσει να τους σταματήσουν όλα αυτά τα στοιχεία που υπήρχαν. Ναι, πρέπει να μιλήσουμε για ευθύνη. Ως πράσινη όμως ξέρω πολύ καλά ότι η πρόκληση της επιβολής προς της ασφάλειας, όσο σοβαρή και αν είναι, δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις. Είχατε τα θέματα του ασύλου, της μετανάστευσης των προσφύγων ως προτεραιότητα ορίσει για την Προεδρία σας. Αυτή οι χωματεροί, αυτοί οι σκυλοπνίχτες που φέρνουν όλο και περισσότερους απελπισμένους από την Ασία και την Αφρική στην Ευρώπη, είναι αυτό που συμβολίζει τα όσα έχουμε κάνει με το Δουβλίνο 1, 2, 3. Είναι αυτά που συμβολίζουν το ότι η Ευρώπη, όσο και αν δεν έχουμε φτάσει στο κατώτερο επίπεδο ε, της κρίσης, γιατί παραμένουμε ένα από τα πιο υψηλά ε, σε εισοδήματα οι πιο ε, σε εισοδήματα χώροι του κόσμου παραμένει ελκυστική για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το παράδειγμα της Ελλάδας έχει να κάνει με, δείχνει μάλλον πόσα λάθη έχουν γίνει σε σχέση με τη σταθεροποίηση και την πολιτική της λιτότητας στην Ευρώπη. Θέλω όμως να πω εκ μέρους της ε, ομάδας μου ότι το ευρώ δεν μπορεί να είναι σταθερό εάν δεν τολμήσει η πολιτική ηγεσία να προχωρήσει στην πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα ή για την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς εδώ δεν έχουμε μπορέσει ακόμη να εξασφαλίσουμε εμπιστοσύνη για μια οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, εκ μέρου τη ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών και, και των Δημοκρατιών τη Ευρώπη, ο κύριο Τσούλο. Πρόεδρε Ρέντζι, πριν από έξι μήνε, αυτή την αίθουσα είπατε ότι αν η Ευρώπη έβγαζε φωτογραφία των εαυτό τη, ένα αυτοπροτέτο, θα βλέπαμε το πρόσωπο τη ανία, τη κόποση και τη παρέπιση. Αυτή ήταν η περιγραφή του δικού σα Ιταλικού εξαμήνου όμω. Και αυτό ήταν το πρόσωπο τη Προεδρία σα. Βλέπουμε ότι σε αυτή την αίθουσα τώρα ε, βρίσκεστε εδώ σε αυτή την αίθουσα σαν να έχετε βγάλει από την τσέπη σα μια συμφωνία για την ευελιξία και ε, Με τι πρώτε συζητήσει όμω που έχουν γίνει φαίνεται ότι οι συμφωνίες ε, που συζητιούνται αφορούν τι ελάχιστε προποθέσει. Δηλαδή μόνο οι επενδύσει που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προωθήσει θα επιτραπούν. Πολύ λίγα σε σχέση με όσα είχατε υποσχεθεί τον περασμένο Ιούλιο λέμε ότι με αυτό ε, το θεατρικό τέχνασμα δεν θα μας εξαπατήσετε πάλι. Το δικό σας ε, εξάμεινο ήταν το εξάμεινο των χαμένων ευκαιριών. Και αυτό το λέω γιατί όταν κανείς αναλαμβάνει τα, είναι ένα τόσο ε, σημαντικού θεσμικού οργάνου πρέπει να τα δώσει όλα. Διότι εάν πάρει την σκητάλη με δύναμη θα παρασύρει τους πάντες. Αλλιώς χάνει χρόνο. Ήταν ε, πάλι μια χαμένη ευκαιρία ο διορισμός ε, της μαθητριάς σας, της ε, κυρίας Μογκερίνη, στα εξωτερικά. Ένα χαρτοφυλάκι που θα μπορούσε να κάνει μια πραγματική διαφορά. Η Μογκερίνη ακόμη δεν κατάφερε να φέρει στη χώρα μας πίσω τους πεζοναύτες. Μια χαμένη ευκαιρία για την ανάπτυξη και την απασχόληση, που τόσο πολύ εσείς ευγελιστήκατε στην αρχή του εξαμήνου. Δεν προτείνεται κανένα συγκεκριμένο μέτρο και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και στην ε, ε, Ιταλία όπου το 43% των νέων είναι χωρίς δουλειά και 13,4% είναι η ανεργία για το σύνολο του πληθυσμού. Χάσαμε την ευκαιρία λοιπόν για τις επιχειρήσεις μας. Μέχρι να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο για το Made in, ούτε αυτό δεν πετύχατε. Συμφωνία που τόσο πολύ σας προσέφερε το Κοινοβούλιο σε ασημένιο αλλά Εσείς το παραμελήσατε. Χαμένες ευκαιρίε όμως κι άλλε για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Ε, ουσιαστικά εξυπηρετήθηκαν μόνο όσοι είχαν μεγάλα συμφέροντα. Ή μετά με τα γάματα φόμικρων, τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, και αυτούς τους ρίξατε για να ωφελήσετε τις πολυεθνικές τη βιοτεχνολογίας. Ή το πρόγραμμα τρίτων, η συγχρηματοδότηση που παραμένει θέμα καλής θέλησης των μεμονωμένων κρατών. Η συμφωνία TTIP που μπορεί να δυσχεράνει συνολικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα για, την, για το ψηφιακό θεματολόγιο δεν προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για να γίνει συγχρονότερη και πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας. Για να γυρίσω λοιπόν στην εικόνα του selfie, του αυτοπορτρέτου που τόσο πολύ σας αρέσει κυρία Ρέντζη, να πω ότι τελικά δεν μπορούμε ε, στην επιφάνεια να κοιτάμε μόνο τα χαμόγελα, γιατί πίσω είμαστε κι εμείς που έχουμε δυσαρεστημένη Ευχαριστώ. Äh, το λόγο έχει ο μη εγγεγραμμένος βουλευτής, κύριος Σαλβίνη. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. το εξάμεινο δεν το οδήγησε σε ε, αποτυχία η Λίγκα του Βορρά, αλλά αυτό το σώμα. Όλοι οι πολίτες που έχουν ε, συνδεθεί στο διαδίκτυο δεν ασχολούνται με το δικό μου πρόσωπο, αλλά με τις κάμερες που έχουμε θα δουν αυτή την αίθουσα και το τι γίνεται. Και θα δουν τα μηδενικά, την έρημο ένα αξιοπρεπές, το τέρμα που αξίζει σε ένα εξάμεινο μόνο λόγια. Το εξάμεινο του κυρίου Ρέντζη, ο οποίος ήρθε εδώ για να ακούσει το μηδενικό που έχει να μας παρουσιάσει και να το εκφωνήσει. Λόγια του αέρα, ε, κάποιο που πριν από έξι μήνες μας έδινε 80 σελίδες υποσχέσεων. Η Ευρώπη θα κάνει μια νέα αρχή, μας είχε πει. Τώρα μας δίνει σελίδες και φύλλα για αυτά που υποτίθεται ότι έγιναν. Και τι έχει γίνει. Ρεκόρ ανεργίας. Λάθος νόμισμα, το ευρώ που κανείς δεν το αφισβητεί. Άμυνα των επιχειρήσεων, μηδέν. Για την άμυνα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τα παραποιημένα προϊόντα της Κίνας, μηδέν για την εργασιακή πολιτική και το τι συμβαίνει με του εργαζομένου στα παραθεριστικά κέντρα, μηδέν. Γεωργική πολιτική, μηδέν. 4.000 ε, ε, εταιρείε παραγωγή ρυζιού, γιατί μα έχει κατακλείσει το ρύζι τη Καμπότζη. Μηδέν. Συμφωνία με το Μαρόκο στο όνομα του διαλόγου και όπου μετατοπίζονται ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και κλείνουν στην Ευρώπη, ενώ άλλε πολυεθνικέ πάνε στην Αφρική. Τέλεια. Ε, βλέπουμε δύο Ευρωπαίοι στρατιώτε από χρόνια να είναι κρατούμενοι στην Ινδία και βλέπουμε να υπάρχει κάμια διάθεση επιστροφή του. Μηδέν. Μεταναστευτική πολιτική έχει αλλάξει το όνομα, αλλά δεν έχει αλλάξει το νόημα. Μπορεί να το ονομάσετε Τρίτονα, Μίκη Μάου ή Πλούτονα αυτό που κάνετε. Αλλά τι θα γίνει με τα εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτεών που απειλούνται. Μηδέν. Η Ρωσία, και για αυτό το θέμα, αντί να πηγαίνετε βόλτε στο Παρίσι, όπου πολύ σωστά κατέβηκαν στου δρόμου τόσοι άνθρωποι, θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογο με τη Ρωσία, που είναι ένα εχθρό κατά του Ισλαμικού εξτρεμισμού. Ένα πράγμα κατά από αυτό το μηδενικό στη σελίδα 11 του προγραμματό σα αναφερόταν η πρόθεση να επανακινηθούν οι διαπραγματεύσει για να μπει η Τουρκία στην Ευρώπη. Ευτυχώς στο μηδενικό σας προστίθεται και η μία έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε, καλή τύχη και ζήτω η Λετωνία που σίγουρα κάτι παραπάνω θα κάνει σε σχέση με την δραματική Ιταλική Προεδρία. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Ρόιλ. Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτού του εξεμήνου το εξέθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Η εξυγίανση των προπολογισμών, η στήριξη των τραπεζών. Βεβαίως μιλούμε για την εμπιστοσύνη του πολίτη και η συνέπεια που προκύπτει τώρα κύριε Προεδρεύων είναι ότι θα πρέπει να ανατραπεί όλη η πολιτική, έτσι λέτε. Εγώ ελπίζω να μην συμβεί αυτό, γιατί αυτό το οποίο έχει κάνει αυτή η πολιτική μέχρι τώρα ήταν μια πολιτική σταθερότητας, εμπιστοσύνης, ανάπτυξης, ότι αυτό που υποσχόμασταν το τηρούσαμε και λαμβάναμε τα μέτρα ένα-ένα, six-pack, two-pack και προχωρούσαμε. Δεν νομίζω ότι κάναμε τόσο άσχημα αν κοιτάξουμε τα αποτελέσματα στην Ισπανία και την Ιρλανδία, Φερρυπίν. Ξέρω ότι σε μια περίπτωση δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα, αλλά τότε θα πρέπει να διερωτηθούμε τι πταίει. Και με αυτό θα πούμε ότι πρέπει να τα ανατρέψουμε όλα, να τα πετάξουμε όλα από το παράθυρο. Όλα αυτά που κάνουν ε, να είναι πιο ασφαλής και πιο σταθερή η οικονομία και οι μεταρρυθμίσεις να προχωρούν, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα τα αναιρέσουν όλα αυτά. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα αποτελέσματα. Εάν ο πολίτης καταλαβαίνει ότι φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα αυτά που κάνουμε και ανάπτυξη, γιατί αυτό δεν θα εξαρτηθεί από το πεστρό χρήμα ή από, από τα ωραία λόγια, αλλά από το αν είμαστε αποφασισμένοι αυτά που υποσχόμαστε να τα τηρούμε. Γι' αυτό και ελπίζω το Συμβούλιο, η Επιτροπή και ε, το Κοινοβούλιο, αλλά και τα κράτη-μέλη να το έχουν αντιληφθεί. Ευχαριστώ πολύ. Mr. there is a blue card for you. Έχετε μπλου κάρτα, κύριε Ρόιλ. Θέλετε να απαντήσετε? Παρακαλώ. Καλή χρονιά. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε αυτά που βλέπουμε από τον κύριο Ρέντσι; τι είναι, είναι μια εικονική παρουσίαση για έναν ιδανικό κόσμο ή συμφωνείτε μαζί του ότι τελικά ο κόσμος αποτελείται από άξες τους οι οποίοι τελικά κάνουν αυτά που κάνουν και εκείνο τελικά δεν ασχολείται με το να βοηθήσει να τα αποφεύγουμε. Απάντηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Εκφράστηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής, υπήρξαν προτάσεις από τον Προεδρεύοντα ότι πρέπει να ανατραπούν τα πάντα. Αυτό το είπα και εγώ, ότι δεν θέλει να κρατήσει τίποτα. Αλλά δεν θα σας ακολουθήσω στο να ε, συμφωνήσω σε ίδρυση βάρος των πολιτικών, γιατί αυτό δεν μας βοηθάει να προχωρήσουμε. Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Γιούνκερ, κύριε Πρωθυπουργέ Ρέντζι, η Ιταλική Προεδρία θα μείνει στη μνήμη μα για μια σειρά από πρωτοβουλίε, ιδίω όσε αφορούν το Ταμείο μια Τραπεζών ή την ε, νομιμοποίηση παράνομου χρήματο. Όμω κυρίω γιατί είχε την τόλμη και την ευθεία να συμπεριλάβει στο πολιτικό θεματολόγιο δύο από τα βασικότερα ζητήματα για την επιβίωση του ευρώ και του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Η συμφιλίωση μεταξύ τη πειθαρχία στα δημοσιονομικά και η εποπτεία για όφελο τη ανάπτυξη και τη απασχόληση, μαζί με τις ε, στατικές επενδύσεις είναι απαραίτητα. Μπορεί να φαίνονται σε κάποιου κοινότοπα, αλλά δεν είναι. Ε, η Ιταλική Προεδρία έφερε στο σύστημα αυτό σοβαρή συζήτηση για τις θεμελιωδέστερε πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώθηκε, άλλαξε. Άλλαξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεφεύγει από το τέλμα με τον κίνδυνο αποπληθωρισμών και την δυσπιστία των Ευρωπαίων πολιτών προς το ευρωπαϊκό εγχήμερο. Στην πραγματικότητα όμως η Ιταλική Προεδρία ακόμη δεν έδωσε την ένεση ζωτικότητας και ενέργειας που χρειαζόταν για να ξεπεράσουμε αυτό το σημείο φάνηκε αδύνατο. Όμως μετά από χρόνια δογματισμού τυφλής λιτότητας και ε, καταπίεσης της ελπίδας, η νέα Επιτροπή Γιούνκερ και η Ιταλική Προεδρία ξεκίνησαν, ξεκίνησαν τουλάχιστον να αγγίζουν τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και να στοχεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ολοκληρώθηκε τίποτα όμως. Άνοιξαν οι πόρτες ξεκίνησε η πορεία για τον δρόμο που πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά που πρέπει να γίνει σε κάθε χώρα και σε συλλογικό επίπεδο. Ε, Βεβαίω, είναι προφανή τα όρια, τα κενά, οι ελλείψει του ευρωπαϊκού οικοδομήματο και κυρίω του κοινού νομίσματο. Όμω, πρέπει η μελέτη μα να συνεχιστεί και πραγματικά εύχομαι η λετωνική προεδρία να μην χάσει λεπτό, αλλά να ευχηθώ ταυτόχρονα ότι η Ιταλία, ε, φεύγοντα από το Συμβούλιο και ω απλό κράτο μέλο πλέον, δεν θα χάσει ρότα τη. Χρειαζόμαστε την Ιταλία στην Ευρώπη. Οι πολίτε που εδώ εκπροσωπούμε πρέπει να ξαναβρούν την ελπίδα του. Πρέπει πάνω απ' όλα να ξαναβρούν την ψυχή τη Ευρώπη. Ευχαριστώ λοιπόν την Ιταλική Προεδρία και ε, πραγματικά να μην ξεχνάμε τον αγώνα για την ελπίδα που έχουμε μπροστά μα. Ευχαριστώ. Ε, Ο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την Ιταλία για την Ιταλική Προεδρία στο Συμβούλιο. Και θέλω επίσης να χρησιμοποιήσω και την ευκαιρία αυτή, κύριε Ρέντσι, προκειμένου να σας ευχαριστήσω επειδή τελικά προχωρήσατε στη στρατηγική Αδριατική Ιωνίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πιστεύω ότι οι χώρες που εμπλέκονται στην στρατηγική Μάλλον πιστεύω ότι θα έχουν ευκαιρία οι χώρες αυτές που εμπλέκονται, Σλοβενία, Ελλάδα, Ιταλία, αλλά και χώρες που βρίσκονται στην περιοχή και που δεν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι δικαίως έχουν πολλές προσδοκίες από τη στρατηγική αυτή όλες αυτές οι χώρες. Οπότε παρακαλώ κύριε Ρέντσι η Ιταλία να παραμείνει υπέρ της στρατηγικής αυτής και τα επόμενα χρόνια. Γιατί αν εσείς δεν φροντίστε για τη στρατηγική αυτή, δεν θα αποκτήσει στρατηγική σάρκα και οστά. Πολλές προσδοκίες υπάρχουν λοιπόν από την στρατηγική αυτή και περιμένουμε ενεργά να συμμετάσχετε στην πραγματοποίηση των όρων της στρατηγικής αυτής κύριε Ρέντσι. Ευχαριστούμε κύριε Φορέντσα. Κύριε Φορέντσα, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω τη μεταφορά του αυτοποτρέτου του Σέλφι. Εγώ θα μιλήσω πιο πολύ για αυτό το πέπλο ρητορίας, διότι με την ε, φωτογραφία αυτή ουσιαστικά χάσαμε την ε, ε, ελπίδα και θα έλεγα να, για το μέλλον και να αφήσουμε λίγο αυτέ τι αυταπάτε και αυτέ τι μεταφορέ για να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Το Τον έχω και τι μελλοντικέ γενιέ αναφέρατε. Και βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η ανεργία των νέων είναι στα υψηλότερα ιστορικά επίπεδα. Ε, εδώ άκουσα πολλά λόγια. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι το πρόγραμμα Juncker. Ευελιξία. Ευελιξία είναι ο σεβασμός των συνθήκων και των συμφώνων σταθερότητας, όπως ακούστηκε εδώ στην Ολομέλεια ή είναι δημοκρατία αυτό που προσπαθείτε να συμπεριλάβετε στο ε, TTIP, στις διαπραγματεύσεις TTIP. Μήπως θα αμυθούν οι νέοι που θα δουλέψουν στην Διεθνή Έκθεση, στην ΕΞΠΟ. Είδατε πόσα εκατομμύρια πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στην Ιταλία για, την, για τις προσλήψεις με επισφαλείς συνθήκες, για την κοινωνική ανεργία. Ακούτε τις φωνές που έρχονται από την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη σκεφτόμενοι ότι θα εξοριστεί από την ήπειρό η Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι η Ελλάδα με την νίκη του Αλέξη Τσίπρα θα ανοίξει το δρόμο για μια Ευρώπη της ελπίδας και για να γίνει το μέλλον που θέλουμε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε κύριο Λαπανσού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ω Γάλλο, θέλω να σα ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σα στην ιστορική πορεία του Παρισιού και πιστεύω ότι είναι σωστοί οι λόγοι οι οποίοι σας οδήγησαν εκεί. Και ευχαριστώ και τον πρόεδρο Γιούγκερ για αυτά που είπε. Συμφωνούμε μαζί σας κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου όταν είπατε ότι τα πιο χρήσιμα που κάνατε για την Ευρώπη είναι οι μεταρρυθμίσεις στην ίδια την Ιταλία. Άλλες κυβερνήσεις της δικιάς μου χώρας για παράδειγμα θα έπρεπε να εμπνευστούν από το θάρρος σας αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στο επίπεδο των υποσχέσεων που δοθήκανε αρχικά. Θα αναφερθώ σε δύο κάπως αφήσιμα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα για τον προπολογισμό. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προπολογισμό για το 2015. Αλλά τα 25 δισεκατομμύρια που είναι απλήρωτοι λογαριασμοί θα εμποδίσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε νέες πολιτικές φέτος. Δεύτερον, ο έλεγχος στη θάλασσα στη Μεσόγειο. Εμείς χαιρετίζουμε την απόδοση και το θάρρος της Ιταλικής ναυτικής δύναμης με το Μάρε Νάστρομ και το τρίτον το οποίο ακολούθησε, αλλά ο τρίτονος δεν έχει χρήματα και κινδυνεύει να είναι λιγότερο αποτελεσματική η πολιτική αυτή για τους ναυαγούς και για να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική πίεση. Έπειτα, το θέμα των πόρων έχει αναβληθεί για αργότερα και αυτό είναι κρίμα. Ευχαριστώ. Κύριε Λαμασούρ, έχετε δύο μπλε κάρτες. Θέλετε να απαντήσετε. Ο κύριος Σκόμπορντ και η κυρία Μούρη, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Uh, Συμφωνείτε μαζί μου ότι η Ιταλική Προεδρία που θα τη θυμόμαστε για δύο πράγματα, την κατάρρευση του ευρώ την δεχόμενη έξοδο από το ευρώ της Ελλάδας και της Ιταλίας και το Wikileaks που βέβαια πλήττει πιστεύω και την Προεδρία. Η ερώτησή σας ποια είναι, ρωτάει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, ο κύριος Μόιε τώρα. Ή όχι. Ναι, κυρία Μόιε. Είπατε ότι η Ιταλική Προεδρία σας ενέπνευσε σας ενέπνευσε και σε αφορά τις απατές τις ατασταλίες της δικής μας πολιτικής τάξης που τόσα χρόνια επιτράπησαν η Διεθνής Έκθεση στο Μιλάνο, η μαφία, οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Δεν κάνατε τίποτα και όλα τα κρύβατε στην επιχείρηση Μόζη, στη Βενετία, εκλάπησαν εκατομμύρια δημόσια και τίποτα δεν υπόθηκε για όλου αυτού του διθαμένου. Κανεί δεν είναι ένοχο και όλοι είναι προστατευμένοι. Στη Ρώμη η μαφία είναι θεσμοθετημένη. Αυτά σα ενέπνευσαν. Μπράβο σα. Ο κύριο Λαμασούρ. Σας ευχαριστώ. Στους δύο ρωτώντες θα έλεγα ότι αντίθετα από αυτούς, εγώ δεν είμαι Ευρωπαίος Φεντεραλιστής. Θεωρώ λοιπόν ότι ό,τι έγινε στην Ελλάδα, ό,τι έγινε στο Λουξεμβούργο, ό,τι έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού δεν είναι πράγματα που εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιταλική Προεδρία, αλλά από την κάθε μία από τις εν λόγω χώρες. Επίσης θα έλεγα γιατί οι κατηγορίες προσάπτεται στην Ιταλική Προεδρία. Δεν είναι εδώ ο χώρος, πρέπει να απευθυνθείτε στον Πρωθυπουργό σα. που βρίσκεται εδώ βέβαια. Ο κύριο Γκουαλτιέρη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω τα λόγια με τα οποία ο πρόεδρο Γιούνκερ εξόρισε την αναγνώρισή του προ τι σημαντικέ αποφάσει του Σώματος Επιτρόπου που πρόκειται τώρα να εγκριθούν, δηλαδή ο κανονισμός για το πρόγραμμα επενδύσεων και ανακοίνωση για την ευελιξία, αυτά είναι πράγματα που επενέπνευσε η Ιταλική Προεδρία. Και αυτό θα πρέπει να μας... αυτά τα θέματα θα πρέπει να κλείσουν τη συζήτηση για τα αποτελέσματα αυτή τη Προεδρίας. Βλέπω εδώ πραγματικά έναν απατηλό και εκφοβιστικό λαϊκισμό να ακούγεται σε αυτήν την αίθουσα και κατά της Ιταλικής Προεδρίας. Υπήρξαν θέματα πολύ μεγάλης σημασίας που ξεπερνούν τα παραδοσιακά ζητήματα που καλύπτουν οι εξαμηνίες Προεδρίας. Ήταν θέματα ουσίας. Παρά τον εκνευρισμό του ε, συναδέλφου Βέμπερ, οι ανακοινώσει θα δείξουν όμως ε, λαμπρός ότι η ευελιξία καλύπτεται από τους κανόνες που θα προταθούν. Η ευελιξία στους κανόνες δεν ε, ε, θα εφαρμοστούν μέχρι τώρα έλειψαν και ε, έτσι ζημιώθηκε μόνο η οικονομία μας. Δεν, δεν είναι αυτός σκοπός οι κανόνες. Στην ε, ε, Ευρώπη θέλουμε την πολιτική και κοινοβουλευτική αναγέννηση της Ευρώπης και στους δρόμους του Παρισιού είδαμε ότι η Ευρώπη δεν είναι απλώς γραφειοκρατία. Αυτό είναι το στίχημα που θέλουμε να ε, νικήσουμε. Η Ευρώπη να έχει πολιτική φύση και νομίζω ότι αυτό είναι η διαρκέστερη νίκη που έχει πετύχει η Ιταλική Προεδρία. Κύριε Γκουαλτιέρη, υπάρχει γαλάζια κάρτα από την ε, κυρία Πιτζότο. Θέλετε να απαντήσετε. 30 δευτερόλεπτα. Οι γαλάζιες κάρτες σκοπό έχουν να θέσετε ερωτήσεις στον ε, τελευταίο παρεμβαίνοντα. Όχι για δική σας παρέμβαση. για, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε. Παρακαλώ, σεβαστείτε τον κανονισμό. Κυρία Μπιτζότο. Κύριε Γκουαλτιέρη, μιλήσατε για τα αποτελέσματα. Στην Αταλία όμως αυξήθηκε η ύφεση, η ανεργία, κλείσαν επιχειρήσεις. Εσείς διαβάσατε, διαβάσατε τα στοιχεία αυτά. Μιλήσατε με πολίτες και επιχειρηματίες. Διότι αυτή την αισιοδοξία που εσείς εκφράσατε και ο πρωθυπουργό μα, ο κ. Ε, δεν, το καταλαβαίνουν οι Ιταλοί. Τα πράγματα απλώ χειροτερεύουν εκεί. Φτάνει λοιπόν αυτές τις αναγγελίες, φτάνει με τα ωραία λόγια, διότι χειροπιαστά τα προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν σε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Κύριε Κουρτιέρη, βλέπω ότι έχουμε περάσει σε ζήτημα τελείω εθνικό. Όμω η Ιταλική οικονομία ε, είναι σε ανησυχητική κατάσταση και επειδή έχουν γίνει λαθασμένε επιλογέ επί πολλά χρόνια. Κυρίω από κυβερνήσει, τι οποίε εσεί και το κόμμα σα δώσατε εμπιστοσύνη από πολλά χρόνια τα χρόνια, ε, ε, αυτό το εξάμεινο μάλλον αντιθέτω, για πρώτη φορά έβαλε τα θεμέλια για μια αλλαγή ε, πορεία και ρότα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Η ανακοίνωση που θα εγκριθεί στη μία μπορεί να μην δώσει αναδρομικά αποτελέσματα για καμία προεδρία νομίζω. Όχι για μα, θα ήταν σούπερμαν όποιο το πετύχαινε αυτό. Αλλά σήμερα τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Το, το Σώμα των Επιτρόπων θα τα εγκρίνει επίση. Αλλάζει η κατεύθυνση συνολικά τη ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό είναι ένα γεγονό που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Είναι ένας, μια διτή επιτυχία τη Ιταλία. Ευχαριστούμε κύριο Φαντελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Ρέντσι για τα όσα κατάφερε αυτό το εξάμεινο. Γιατί είχατε ένα φιλόδοξο θεματολόγιο σε μια εποχή όπου η οικονομική κρίση έπλητε αδυσόπιτα το δυτικό κόσμο. Έχετε, αναλάβατε μια προεδρία με νέο κοινοβούλιο και νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως Ξέρουμε πάντα ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και να έχουν γίνει και περισσότερα και σε αυτό θα συμφωνήσω. Όπω είπε και ο κύριο Γκίφερ Χόφστα, το ηγέτη τη ε, πολιτική μου ομάδα, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα για το πακέτο των τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, ένα άλλο θέμα στο οποίο θα έπρεπε να έχουμε ε, ω Ευρώπη επιδιώξει περισσότερο ήταν η κλιματική στόχη, όπου κατέβασε το επίπεδο των προσδοκιών και απαιτήσεων το Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι χάνουμε τόσο την ευκαιρία των επενδύσεων όσο και το βηματισμό μας σε σχέση με το μέλλον γιατί θα χρειαστεί αργότερα να επιταχύνουμε σημαντικά για να καλύψουμε ε, προθεσμίες, όρια και στόχους που θα έπρεπε ήδη να έχουμε ξεκινήσει να επιδιώκουμε. Κύριε Φέντερλη, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας διατεθειμένος να τη δεχθείτε. Γκραντίνη παρακαλώ. Γκαρντίνη μάλλον. Γκραντίνη, γκραπίνη και όχι γκαρντίνη. Η κυρία Γκαρπίνη. Γκραπίνη. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είπατε κύριε Σνάλφα ότι για το περιβάλλον η Επιτροπή μας οδήγησε σε απογοήτευση. Νομίζω ότι δεν ήταν αυτός ο μόνος τομέας. Ε, πιστεύετε ότι μπορούν με κάποιες τροποποιήσεις να βελτιωθούν οι προτάσεις της Επιτροπής απάντηση. Ναι, βεβαίως πάντοτε είμαι διατεθειμένος να επιδιώκω πρόοδο όσον αφορά την πράσινη πολιτική. Γιατί είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το μέλλον της Ευρώπης ανήκει στην πράσινη οικονομία για θέσει εργασία και και επενδύσει. Καθώ όμω δεν μιλούσαμε για το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά για την Ιταλική Προεδρία, είχα σημειώσει ότι πολλά ακόμα θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά πολλά έχουν και επιτευχθεί. Και ότι ήταν οι συνθήκε δύσκολε με νέο κοινοβούλιο, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αδυσόπιτη οικονομική κρίση. Χωρί αυτό να σημαίνει δεν μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερο, να επιδιώξουμε από εδώ και προ περισσότερα προ την κατεύθυνση τη πράσινη οικονομία. Κυρία Γκαρντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πρέπει να πω ότι δεν φτάνει η καλή πρόθεση που μπορεί να έχουμε Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα μεγάλος ενθουσιασμό. Κάτι λίγο πιο χειροπιαστό θέλαμε. Μετά από τόσα χρόνια που είμαστε στην Ευρώπη. Και εμεί οι Ιταλοί ε, έχουμε συνηθίσει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Διότι όλοι περιμένουν να περάσουμε στην ουσία των θεμάτων. Τώρα, εάν έχουμε ανοίξει μια γραμμή πίστοση, όταν είπαμε για ανοίγματα, με τόσα ωραία λόγια και δόθηκαν τόσε υποσχέσει, και λέτε ότι θα περάσουμε στη μελλοντική και μελλοντολογική Ευρώπη σήμερα, αυτή η όθηση τη Ευρώπη ε, που κοιτάζει προ το μέλλον, είναι λίγο εκτό θέματο. Εδώ απολογισμό θέλαμε να κάνουμε. Ε, ήταν ωραίο να ρίξουμε ίσω την τράπουλα για να δούμε τι θα γίνει, τα χαρτιά, αλλά, ε, να διαβάσουμε τα ταρό, αλλά δεν είναι αυτό ο στόχο εδώ. Ε, ο στόχο του Ιταλικού εξαμήνου που φτάνει σε ένα τέρμα σήμερα ήταν να δούμε τι κάνατε και δεν ήταν ε, κάτι που μα ενθουσιάζει ο απολογισμό. Κάτι πιο χειροπιαστό θέλαμε για τα θέματα που μα απασχόλησαν, θέματα που δεν θα διακόπουν βέβαια, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άκοπα γι' αυτά, θεωρώντα ότι είναι θέματα σημαντικά για τους συμπολίτε μας, αλλά περιμένουμε τουλάχιστον κάτι παραπάνω, κάτι για την οικονομία, για την ανάπτυξη. Μιλήσατε για το Μεντίν, μιλήσατε για τόσα πράγματα που δεν έχουν λάβει σάρκα και ωστά αλλά δεν είπατε τίποτα δεν είπατε πώ θα αντιμετωπίσουμε την κατεπίγουσα ανάγκη αυτών των τελευταίων ωρών. Η επιχείρηση Τρίτονα, τι στάση θα πρέπει να έχει όμως η Ευρώπη απέναντι στο Ισλαμικό κράτος που έχει γίνει ε, ένα οχυρό για όλους τους εξτρεμιστές Ισλαμιστές όλου του κόσμου. Με το σύμφωνο σταθερότητας επίσης. Ε, αυτό ήταν κάτι που μπορούσε να λυθεί έτσι κι σε λίγες ώρες. Το μεγάλο θέμα με το οποίο ξεκινήσατε το ταξίδι σας πριν από έξι μήνες ήταν λιγάκι αυτό ε, το παιδάκι, η εικόνα του παιδιού που βλέπει τη μητέρα του να κάνει το κλασικό νοικοκυριό και να απασχολείται στο σπίτι, ενώ περιμένει νέα από χρόνια που τελικά δεν έρχονται ποτέ. Αυτή την εντύπωση μα δώσατε στο εξάμεινο τη Ιταλική Προεδρία. Πρόεδρο, παρακαλώ, ε, αν μπορούμε, μία γαλάζια κάρτα αναπαράμβαση για να. Και επίσης να περιορίζεστε αν γίνεται σε ερωτήσεις κάθε φορά. Κυρία Γκαρντίνη, θα απαντήσετε στην ερώτηση της κυρίας Μπρέσο. Κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα θέλω απλώς να ρωτήσω την κυρία Καρδίνη. Εδώ λέμε και ξαναλέμε ότι πρωταρχικός μας στόχος είναι η Ευρώπη να επιστρέψει σε ρυθμό ανάπτυξης και ανάπτυξη ίσων επενδύσεις. Εδώ έχουμε δύο αποτελέσματα, όχι μόνο του προγράμματος Juncker, αλλά και της δυνατότητας μέσω του χρυσού κανόνα να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν επενδύσεις απευθείας ε, είναι σημαντικότερα, σημαντικότερα τα στοιχεία αυτά. Δεν θεωρείται ότι αυτά είναι χειροπιαστά αποτελέσματα. Οι άλλοι ανέφεραν διαφορετικά πράγματα. Δεν έχω εδώ χρόνο να τα πω όλα, αλλά τα βρίσκω πολύ χειροπιαστά. Ιδίω στην αυστηρή γραμμή ε, των όσων καταφέραμε αυτού του λίγου μήνε που είχαμε την Προεδρία, αλλά είχαν ήδη ζητηθεί ει και στο παρελθόν η ε, κυρία Γκραντίνη. Κοιτάξτε, επ' αυτού νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτω ή άλλω. Χαίρομαι, χαίρομαι που η Ιταλική Προεδρία, όπω θύμισε και ο πρόεδρο Γιούνκερ, που συνεργάστηκε και δεν παρεμπόδισε το έργο τη Προεδρία προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά κατεύθυνση αυτή γιατί ε, ήταν κάτι που το ΕΛΚ το είχε ζητήσει από την περασμένη άνοιξη στη Σύνοδο του Δουβλίνου πολύ πριν την Ιταλική Προεδρία. Συνεχίσαμε, εντάξει, αλλά χειροπιαστό. Ήθελα να πω πώ ακριβώ θα λάβει αρκετά και ε, όλη αυτή η ωραία ομιλία στην Ιταλία, για το οποίο δεν ξέρουμε τίποτα. Μίλησε ο Πρωθυπουργό. Ε, ο πρόεδρο του Συμβουλίου, ενώ δεν μίλησε καθόλου για αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε, κύριο Λέκφιν. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ. αναλάβατε την Προεδρία σε ταραγμένες εποχές και χρειάστηκε να, να, αντιμετωπίσετε τους ανέμους που έπνεαν. Υπάρχουν λοιπόν δύο αντιδράσεις του ναυτικού όταν πνέει ο άνεμος δυνατά. Είτε πάει και κρύβεται, είτε ακολουθεί και αντιμετωπίζει τον άνεμο και τις συνθήκες. Αυτό μπορέσατε να κάνετε, αυτό επιλέξατε να κάνετε, ήταν σκληρή η δουλειά. Μπορέσατε να διαπραγματευτείτε για τα λεγόμενα gigaliner, τα πολύ μεγάλα φορτηγά. Μπορέσατε να αντιμετωπίσετε ένα μεγάλο πακέτο με μια μεγάλη λύση ικανοποιητική για όλους. Πολύ καλά. Αυτό πρέπει να το καταδείξουμε ως επιτυχία της Προεδρίας σας και δεν καταλαβαίνω τους συναδέλφους οι οποίοι ούτε καν συμμετέχουν στη δουλειά αυτή, που πάντα καταγγέλουν, που πάντα είναι ε, αντί, ενάντι, αντίπαλοι, αλλά δεν βοηθούν να αλλάξει τίποτα. Αυτά λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι είναι απλώς διπλό Η κυρία Βίκστρομ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλω να υποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να ευχαριστήσω την Ιταλική Προεδρία για το εξαίρετο έργο τη στου διάφορου τομεί με του οποίου ασχολήθηκε. Μετά όσα έγιναν τι τελευταίε μέρε στη Γαλλία, δεν έχει νόημα να συζητάμε για το Μεντίν, για παράδειγμα. Το Μεντίν μας φαίνεται δευτερεύον. Καλό είναι να συζητάμε για τις διάφορες προδιαγραφές, αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι τα ουσιώδη. Το θέμα λοιπόν των σημάτων στην Ευρώπη είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ξέρετε ότι έχω δουλέψει μαζί διπλωμάτες του επίπεδου για χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι τελικά χάρη στη δικιά σας προετοιμασία θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την υπόθεση αυτή. Η Ευρώπη των πολιτών πρέπει να ενισχυθεί και ενισχύεται βέβαια όταν υπάρχει αυτός ο πόνος όπως είδαμε με την πορεία της Κυριακής. Πρέπει να περισχύσει η ελευθερία έκφρασης, η διαφάνεια. Τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθος στην Ευρώπη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να πιστέψουμε και να είμαστε πιο επιθετικοί σε ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω διάφορα προβλήματα αλλά και διάφορα θέματα τα οποία οδήγησαν στην επιτυχία της Ιταλικής Προεδρίας. Οικονομικά μιλώντας μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος Ρέντσι τα κατάφερε αρκετά καλά. Οδηγηθήκαμε σε συμπεριφορές που οδήγησαν και πάλι στην αρχή της ανάπτυξης και θέλω τώρα να έρθω στην Ισπανία. Επιτρέψτε μου. Το σχέδιο Juncker έχει φέρει ελπίδα βέβαια για το μέλλον. Και θέλω επίσης να πω ότι πετύχαμε μια καλή ισορροπία. Στην εξωτερική πολιτική πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε τη θέση την οποία έχει και θα έχει κατάσταση είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μετά μάλιστα από τις τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσει το PNR, η ανταλλαγή ονομάτων επιβατών. Για τις ελευθερίες μας πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ασφάλειας. Η ασφάλεια δεν είναι θεμελιώδης δικαίωμα. Είναι ένα νομικό κεκτημένο που είναι αναγκαίο και απαραίτητο για να πετύχουμε την ελευθερία και τη διασφάλισή τη. Ευχαριστώ. Η κυρία Σανάλοβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Οι έξι μήνες της τελικής Προεδρίας χαρακτηρίζονται από αλλαγή ε, προσώπων στη, στα θεσμικά όργανα, εκλογή του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκλογή γιουνκερ και της νέας ηγετικής ομάδας της Επιτροπής. Η Προεδρία μπόρεσε να ε, διαχειριστεί τη μετάβαση αυτή ανάμεσα σε δύο θητείες, να προσαρμοστεί αλλά και να ολοκληρώσει τη δουλειά που δεν είχαν ε, κλείσει προηγούμενες προεδρίες. Εγώ ήμουν ε, εισηγήτρια για το σύστημα του ηλεκτρονικού της ηλεκτρονικής ανάγκης ή κόλλ. επίγουσας ανάγκης, η Ε, έχω να διαπιστώσω ότι ήταν πολύ επικοδομητική η στάση της Ιταλικής Προεδρίας και χάρη και στη συνεργασία των Ιταλών συναδέλφων μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε ένα κείμενο το οποίο θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια. Θέλω λοιπόν ρητά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου κύριε Πρωθυπουργέ σε εσά και του συναδέλφου σα. Ευχαριστώ. Γκάμπριελ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Μετά από την Ιταλική Προεδρία νομίζω ότι μπορούμε να σας συγχαρούμε για μια επιτυχημένη θεσμική μετάβαση μεταξύ δύο επιτροπών με διαφορετικό δημοκρατικό εύρος. Αυτή η μετάβαση δίνει νέες πολιτικές προτεραιότητες. Τέσσερις θα αναφέρω. Πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω την υιοθέτηση των συμπερισμάτων όσον αφορά τις μεταστευτικές ώρες και το ξεκίνημα της διαδικασίας του, Καρτούμ, του Χαρτούμ δηλαδή, με τις χώρες του κέρατος της Αφρικής. Είναι μια καλή συνέργεια, είναι μια καλή κατεύθυνση για μια πραγματική διπλωματία της μετανάστευσης. Όμως είμαι πολύ πιο επιφυλακτική όταν πρόκειται για το τρίτονα και για τα μέσα τα οποία διαθέτει προκειμένου να πετύχει μια αλληλέγγυα πολιτική και αποτελεσματική πολιτική όσον αφορά τώρα τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Διαπιστώνω ότι οι πύλες του Σέγγεν εξακολουθούν να είναι κλειστές για την Βουλγαρία και την Ρουμανία, παρά την τήρηση των τεχνικών κριτηρίων. Τρίτον, είδαμε τι έγινε με το South Stream. Η ενεργειακή πολιτική πρέπει σήμερα να γίνει αντιληπτή σαν ένα στοιχείο περιφερειακής ένταξης που θα επιτρέψει σε χώρες όπως η Βουλγαρία να συνεχίσουν να στηρίζουν το ευρωπαϊκό σχέδιο και ανοίγοντα προοπτικές και για τις δύο πλευρές και κυρίως για τις χώρες του Νότου. Συγχαίρω λοιπόν την Ιταλική Προεδρία για την διπουργική διάσκεψη που έγινε στην Ρώμη τον Εύρο που μας πέρασε με τις χώρες Euromed. Και λυπούμε που η Προεδρία αυτή δεν κατάφερε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο για διάφορα νομοθετικά ε, σχέδια όσον αφορά την ισότητα ε, ανδρών και γυναικών των Women on Board. Ελπίζω να αλλάξει αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταραβέλα. Κύριε Πρόεδρε, όπως υπογραμμίσε και ο Πρόεδρος Γιούνκερ, μπορέσατε να κλείσετε τους προπολογισμού για το 2014-2015. Επίσης υπογραμμίζουμε τη βούλησή σας για ε, νέα όθηση στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη. Ωστόσο είχατε δύο μενεκτήματα που έχουν να κάνουν με το χρονοδιάγραμμα. Αυτό το ε, πρώτο που συναντούμε κάθε χρόνο, κάθε πενταετία, δηλαδή την ανανέωση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου αντίστοιχα κύριε Ιούνκερ όπου σαν συνέπεια υποφέρει η παραγωγικότητά μας η νομοθετική και δεύτερο μειονέκτημα που πλήττει κάθε προεδρία του δεύτερου εξαμήνου που αναλαμβάνει καθήκοντα την ώρα που μπαίνουμε στις θερινές διακοπές με δύο μήνες έστω όχι απόλυτης αδράνειας αλλά πάντως ε, χαλάρωσης έστω και αν ο πρώτος μήνας ο Ιούλιος έχει αρκετή δουλειά και έτσι θα πρότεινα να αλλάξουν ε, ε, τα χρονοδιαγράμματα των ε, Προεδριών ώστε να πάμε από 1η Φεβρουαρίου και 1η Αυγούστου να ξεκινάνε τη δουλειά του οι Προεδρίε. Είναι μοιρασμένο αυτό το μειονέκτημα. Ευχαριστώ, Σαλίνη. Ευχαριστώ. Είναι πρώτη φορά που είμαι βουλευτή, κύριε Πρόεδρε. Έχοντα ακούσει τη συζήτηση αυτή, έχω την εντύπωση ότι πολλά από αυτά που υπόθηκαν θα τα είχατε πει έτσι κι αλλιώ ε, με την ομιλία σα αυτή δηλαδή κάτι θα έκανε η Ιταλική Προεδρία αλλά δεν έκανε και τίποτα. Και αυτό πραγματικά με στενοχωρεί διότι κάνει τη συζήτηση απογοητευτική και τα, θεμικά επικριτικά, τα θεμητά επικριτικά σχόλια που θα μπορούσαν να ακουστούν τελικά δεν εμπλωτίζουν τη συζήτησή μα. Μιλήσαμε για ένα επενδυτικό πρόγραμμα με περισσότερα από 300 δι. Εντάξει είναι ένα γεγονό. θα είναι κάτι το θετικό γιατί θα ήταν χειρότερο να μην το είχαμε. Ε, ξεκινά από αυτό το ταπεινό στοιχείο. Όμω, κάποιε σκέψει επί τη ουσία με ένα πρόγραμμα πρόγραμμα που έχει και θετικά στοιχεία αλλά και αδυναμίε, είναι σημαντικό το τι θα γίνει με τη μόχλευση λόγου χάρη. Ε, το κατά πόσον στο ε, πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν πολλέ επενδύσει που θα μπορούσαν να είναι στατικικέ αλλά δεν παράγουν τόση κερδοφορία όπω οι επενδύσει των τομέων των συνδρομικών. Ε, εδώ λοιπόν, εφόσον ε, θέλουμε να ασχοληθούμε χειροπιαστά με τα προβλήματα, να πάμε στην ουσία των προβλημάτων, με αυτή τη μεγάλη ελπίδα να χτίσουμε μια Ευρώπη που δεν θα είναι αντικείμενο απλώ συζητήσεων και κενών λόγων, αλλά θέλουμε να αναπτυχθεί και να επιτρέψει στι οικογένειε και τι επιχειρήσει να προχωρήσουν. Αυτή την ελπίδα πιστεύω ότι όλοι τη συμμεριζόμαστε. Όμω στην αίθουσα αυτή πολλέ φορέ ε, βλέπουμε να μην είναι εδώ αυτοί που την κατηγορούν την αίθουσα ότι είναι άδεια, γιατί είναι άδεια αυτή τη στιγμή, αλλά αυτοί που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή έχουν διάθεση να εργαστούν και να μελετήσουν. Η πρότασή μα έχει πολύ σαφεί ρίζε. Θέλουμε ε, ιδεοχριστιανικέ ε, ρίζε και αξίε για την Ευρώπη μα. Αυτέ δέχτηκαν επιθέση και να μην περιμένουμε και άλλα σημάδια συναγερμού. Να εργαστούμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ όλου για τη συνεργασία. Κύριε Σαλίνη, υπάρχει γαλάζια κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε. Από τον κύριο Βάλλη. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσετε το λόγο μετά την τρίτη μου γαλάζια κάρτα που δεν την είχατε δει ίσως, δεν την είχατε ακούσει. Να ρωτήσω τον κύριο Σαλίνη, εφόσον είναι καινούριο. Αλλά συμμετέχει σε ένα κόμμα που εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει λησαλέα το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Όσα πέτυχε ο πρόεδρο Ρέντζε αυτή τη στιγμή για την μετατροπή του ε, Δημοσιονομικού Συμφώνου και του Συμφώνου Ανάπτυξη και Σταθερότητα, πιστεύετε ότι είναι πράγματα που μπορούν δημοσιονομικά να τα αντέξουν οι Ιταλοί. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Θεωρείτε ότι είναι βιώσιμε αυτέ οι λύσει. Τι θα πρέπει να κάνουν τα επόμενα χρόνια. Κύριε Σαλήνη, έχετε το λόγο. Είμαι πεπισμένο για το εξή. Και ω ε, δήμαρχο ε, και πρόεδρο περιφέρεια την ουσία του συμφώνου την έχω ζήσει στο πετσί μου. Δεν μα εμποδίζει να υπάρξουμε το Σύμφωνο Σταθερότητα σε όσου δεν έχουν εναλλακτικέ λύσει για τη δημοσία διοίκηση δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν η αναθεώρηση του κανονισμού για το πρόγραμμα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε έτσι σήμερα. Ζητήσαμε όχι να αποφύγουμε το Σύμφωνο Σταθερότητα, να το αναθεωρήσουμε, να βρούμε μια νέα αντίληψη γι' αυτό. Έχουμε ανησυχίε όπω όλοι, αλλά ε, εδώ η ισχύ εν τη ενώση, δηλαδή με μια χειροπιαστή πρόταση μπορούμε να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, είναι στη διακριτική ευκαιρία τη Προεδρία να δώσει το δικαίωμα γαλάζια κάρτα. Επειδή στην ομάδα σα έχουν γίνει περισσότερε ερωτήσει μέσω γαλάζια κάρτα, σήμερα θα, τη φάση δεν θα σα ξαναδώσω το δικαίωμα ε, για γαλάζια κάρτα ξανά. Ο κύριο Ντάντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, Πρόεδρε Γιούνκερ το εξάμεινο της Ιταλικής Προεδρίας που μόλις έληξε ήταν μια πρώτη, ένα πρώτο δείγμα καμπή στην αλλαγή για την ευρωπαϊκή πολιτική με ευφυείς τροποποιήσεις στις επενδύσεις και την ανάπτυξη της, του ευρωπαϊκού θεματολογίου που πέρασαν πλέον μεταξύ των πολιτικών μας προτεραιοτήτων. Η Μεσόγειος με τα ιταλικά σκάφη βλέπουμε να είναι ένα σταυροδρόμι και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και από τις εκλογές του Μαΐου αλλά αποφασιστική ήταν η στροφή που έκανε η Ιταλική Προεδρία. Προσπαθούμε να μετατρέψουμε λοιπόν αυτή την Ιταλική αλλαγή σε μια συνιστόσα τη Ευρώπη που θα μα επιτρέψει να έχουμε περισσότερο κύρο ω Ένωση στον κόσμο, με περισσότερη προστασία στι κοινωνίε μα και μια ανάπτυξη που να βασίζεται στην πραγματική οικονομία. Τι ημέρε αυτέ είδαμε να ακούγεται πολλέ φορέ ότι περισσότερη Ευρώπη χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τι μελλοντικέ προκλήσει. Θα ήθελα κύριοι Πρόεδροι, εικόνα από την Κυριακή όλοι είδαμε ε, στο Παρίσι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να βαδίζουν ενωμένοι να μεταφραστεί και σε πολιτική δράση. Και ο Αλτιέρο Σπινέλη μα το είχε πει. Ο δρόμο θα πρέπει να κάνουμε δεν είναι απλώς ούτε ασφαλή, αλλά θα πρέπει να τον διατρέξουμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριε Συναδελφέ, όταν αξιολογούμε την ε, Ιταλική Προεδρία, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το τελευταίο εξάμεινο ήταν κατά πάσα πιθανότητα αυτό με τι περισσότερε προκλήσει από την ε, προοπτική τη εξωτερική πολιτική. Από τη ρωσική επέμβαση στην ε, Ουκρανία έως την ανάδειξη της ισχύω του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ ε, είχαμε τεράστιες προκλήσεις και χρειάστηκε να συμφωνήσουμε και τα καταφέραμε σε κυρώσεις ε, από πλευράς της Ευρώπης για την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από πλευράς της Ρωσίας. Τα καταφέραμε λοιπόν εκεί και αυτό είναι σημαντικό επίτευγμα για την κοινή μας πολιτική. Είχαμε αρκετά κράτη-μέλη περιλαμβανομένης της Ιταλίας ταυτόχρονα τα οποία ενώθηκαν στην παγκόσμια στη διεθνή συμμαχία κατά του ISIS ε, για να καταπολεμήσουν την προέλασή του. Επίσης έδωσε ανταπόκριση στην μεγάλη μεγάλη κρίση της μετανάστευσης στη Μεσόγειο με την επιχείρηση τρίτων η Ιταλία. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορεί να μας καθησυχάσει το γεγονός ότι τόσο στην νότια όσο και στην ανατολική γειτονία μας τα πράγματα φαίνονται κάπως πιο σταθεροποιημένα σε σχέση με το καλοκαίρι. Έχουμε αποφύγει και αποτρέψει τα χειρότερα, τις χειρότερες εξελίξεις και αυτό το οφείλουμε στην Ιταλική Προεδρία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Τώρα περνάμε για πέντε λεπτά στη διαδικασία του Καρστιά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν στήσει το λόγο και θα δώσω το λόγο μόνο στου πρώτου από κάθε ομάδα που ζήτησαν να παρέμβουν. Άρα ξεκινούμε με τον κύριο Γιούρεκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εχθές και σήμερα. Ακούσαμε πολλά ωραία λόγια για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όταν όμως χρειάστηκαν αλληλεγγύη οι γεωργοί μας, οι αγρότες μας, όταν τους έπληξε τόσο σκληρά το εμπάργκο κατά της Ρωσίας, ξεχάστηκε, στέρευσε η αλληλεγγύη. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, τα κράτη-μέλη πρέπει να ορθώνει το ανάστημα κατά τρόπο ειρηνικό για την, για την ασφάλειά μας και πρέπει να χαράξουμε έναν δρόμο ουσιαστικό για την ελληνική. Έτσι λοιπόν στο μέλλον όταν θα κληθούμε να αξιολογήσουμε μια προεδρία θα πρέπει και να είμαστε προετοιμασμένοι να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε για να ενισχυθεί η ασφάλεια της Υπήρου μας και να επιδείξουμε αλληλεγγύη προς τους φίλους μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα έχει το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε Ρέντσι, το εξάμεινο της Ιταλικής Προεδρίας είχε ένα καθοριστικό πολιτικό ρόλο σε ένα χρόνο που άλλαξε η νομοθεσία και αναθεωρήθηκε και η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Δίνοντας έμφαση στην πολιτική για τις επενδύσεις, όπως το επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, εφόσον το ενέπνευσε και όχι απλώς ε, επέτρεψε με τη συνεργασία του Ιταλική Προεδρία να επιτευχθεί και την ευελιξία. Ένα σημαντικό τρίγωρο. Έρευνα ε, και ανατομία, ε, τηλεοπτικοακουστικά και πολιτισμό. Αυτό, ε, ξέρετε, Πρόεδρε, ότι στην Επιτροπή Πολιτισμού το επεξεργαστήκαμε με θαυμάσιο τρόπο, χάρη στην Ιταλική Προεδρία και για την νεολαία και για τον πολιτισμό και για τον, τον αθλητισμό και του νέου. Εδώ βλέπετε ότι σημαντικά αποτελέσματα με την εκπαίδευση ως μία από τις πέντε προτεραιότητες του επενδυτικού προγράμματος ε, να δοθεί μεγάλη προσοχή. Η διασύνδεση της ε, η κατεύθυνση της Ένωσης με νέες αρμοδιότητες για την εκπαίδευση και νέες ευκαιρίες εργασίας, χάρη και στην ε, όθηση που έδωσε η δική σας Προεδρία και με τη δική μας δουλειά, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να ελπίζουμε ανάκαμψη και επενδύσεις στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και την, ε, την ευκαιρία και στον πολιτιστικό τουρισμό να δοθούν δυνατότητε και σε προοπτικέ νέα οικονομική ανάπτυξη. Διότι αναθεωρήθηκε και η, Ευρώπη, η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Γι' αυτά σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Παλώμα Λόπε Δεμέχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή σα μέρα. Στην Ιταλική Προεδρία μιλήσαμε πολύ για την ταυτότητα, για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μια ταυτότητα η οποία αποτελείται βέβαια από ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται μεταξύ άλλων στον κοινωνικό διάλογο και στη σημασία που έχουν οι συλλογικέ συμβάσει και διαπραγματεύσει με εργασιακέ συνθήκε που να βασίζονται στο εργασιακό δίκαιο. Τελικά όμω στην Προεδρία αυτή είδαμε για άλλη μια φορά πώ γίνονται μεταρρυθμίσει οι οποίε διαλύουν τι βασικέ δομέ της κοινωνικής προστασίας και της εργασιακής προστασίας και στην Ιταλία, όπως έγινε νωρίτερα στην Ισπανία και αλλού. Δεν δούλεψε η Προεδρία αυτή για οικονομική ανάπτυξη, για απασχόληση. Έχουμε λοιπόν λίγες ε, ελπίδες και προσδοκίες από το σχέδιο Juncker. Αναφερθήκατε στον Οδυσσέα. Ναι, ε, στην Οδύση όμως υπάρχει και η Πινελόπη, η οποία κεντάει και ξυλώνει συνέχεια το, αυτό που φτιάχνει. Συνεπώς αυτό κάνατε κι εσείς. Διαλύσατε το κοινωνικό ιστό της Ευρώπης και αυτές είναι οι βάσεις για να χάσουμε τελικά και την ευρωπαϊκή ταυτότητα για την οποία μιλήσατε. Πρέπει να υπάρχει ελπίδα για αλλαγή μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ευχόμαστε και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. La parola Castaldo. Ευχαριστούμε κύριος Καστάλντο. Πρόεδρε, Πρόεδρε Ρέντσε, ακούσαμε ένα σουρεαλιστικό λόγο σήμερα σε μια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα. Λέτε για μια Ευρώπη που άλλαξε πορεία, μια νέα πορεία για την ανάπτυξη και την ευελιξία με ευρωπαϊκό όραμα. Μα για ποιο όραμα αλλαγή, μιλάτε, Πρόεδρε, αυτό των ανύπαρτων ευρωομολόγων και τα δισεκατομμύρια που έχει υποσχεθεί η Επιτροπή και τον δούριο ύπο που για πολλωστή φορά βλέπουμε να παρουσιάζεται στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών, με το ελάχιστο και υποχρεωτικό εισόδημα γειτονία για την Ήπειρο που δεν υπάρχει με την έλλειψη ζωή, την αποσιώπηση των κοινωνικών πολιτικών στην Ευρώπη. Ε, οι νέε γενιέ στην Ιταλία και σε πολλέ άλλε χώρε έχουν ε, χάσει τα φτερά του, του έχουν κόψει τα πόδια. Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει οδηγήσει σε οικουμενική ανεργία. Όλα αυτά παραμένουν λόγια. Ε, η νεολαία τη Νότια Ευρώπη δεν έχει ελπίδε. Και εδώ δεν του κλέψατε απλώ ένα όνειρο από το σιρτάρι του, κύριε Πρόεδρε, αλλά ολόκληρο το γραφείο του, πήρατε και φύγατε. Εδώ λοιπόν ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον ε, Βορρά που προστατεύει ακόμη το κοινωνικό κράτο, ενώ ο Νότο έχει παραδοθεί στι ε, λησαλέ στις πολιτικέ. αντικοινωνικές πολιτικές. Εδώ λοιπόν όσοι λαιλατούσαν τα σούπερ μάρκετ γιατί δεν είχαν να φάνε, δεν χρειάζονται εδώ τι υποσχέσει μα χρειάζονται τόλμη και παρεμβάσει. Αυτή θα έπρεπε να είναι η Ευρώπη και αυτή είναι η Ιταλία. Ευχαριστούμε ο κύριος Μποργέτσιο. Ο πρόεδρος ε, του εξάμεινου, ε, του, ο προεδρεύων Συμβουλίου, ο κύριος Ρέντσι, μας είχε κάνει πολλές υποσχέσεις για τις επιχειρήσεις. Την κράτησε την υποσχέση του. Ουσιαστικά εξασφάλισε την πτώχευση της επιχειρήσης του πατέρα του με τα δημόσια κονδύλια, ενώ οι μικροεπιχειρηματίες στην Ιταλία αυτοκτονούν ε, απελπισμένοι με τους εργαζομένους τους το ίδιο. Ακούμε καθημερινά εκκλήσεις και μόλις έφτασε στα χέρια μας έκκληση από επιχειρηματίες μικροεργαζομένους της χώρας μας που δεν ξέρουν τι να κάνουν με τις δουλειές τους. Ε, πρόεδρε Ρέντζη, Είσαστε πρόεδρος της κυβέρνησης, αλλά πάψτε να κοροϊδεύετε τις επιχειρήσεις πλέον. Αν θέλετε, αναλάβετε δέσμευση για να, θέσετε θέσεις, για να σώσετε θέσεις εργασίας. Να λύσετε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Κάντε για τους άλλους αυτό που κάνετε και για την επιχειρήση του πατέρα σας που ήταν ε, να πτωχεύσει. Εάν ε, δεν ήσασταν ο πρόεδρος της κυβέρνησης και ο πρωτεργάτης αυτής της Ευρώπης, θα την είχατε χάσει. Ευχαριστούμε. Για να απαντήσει εξ ονόματος του Συμβουλίου ο πρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης, ο κ. Ρέντσι. Ευχαριστώ πρόεδρε Ταγιάννη. Τρία είναι τα βασικά θέματα που μας απασχόλησαν στη συζήτησή μας. Πρώτα απ' όλα ο τεχνικός εννοούμενος απολογισμός της Ιταλικής Προεδρίας. Πραγματικά ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υπογράμμισαν στοιχεία που εγώ ίδιο δεν είχα παρεθμίσει καλά-καλά ε, συγκεκριμένα. Γιατί σα παρέπεμψα στο συμπληρωματικό κείμενο. Όμως ευχαριστώ πολύ για τα λόγια ευχαριστίας και τα σχόλιά σας για τον απολογισμό της Προεδρίας μας, για θετικά στοιχεία που καταφέραμε σε αυτό το εξάμεινο και παραδόξω τα αναφέρατε εσείς στο κοινό και όχι εγώ. Όμω, να πω ότι έχει δίκιο και ο κ. Φερχόφτατ όταν εντοπίζει κάποια στοιχεία που ήταν μη θετικά. Όχι απλώς δεν ολοκληρώσαμε το θέμα του Μεϊντίν, ένα θέμα που θα συνεχίσει να μας απασχολεί, επί το οποίο θα εργαστούμε και για μας είναι ένα στοιχείο αντικειμενικά αρνητικό, αλλά υπάρχει και το θέμα των επικοινωνιών. Πολύ περίπλοκο συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων. 11 φορές συναντήθηκαν οι ομάδες εργασίες με ενδελεχέστατες συζητήσεις που τους παρακολούθησε και το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών στο Μιλάνο με δύο σχέδια κειμένων να έχουν προταθεί και με μερικά βήματα πρόοδου όπως την ε, ουδετερότητα του δικτύου αλλά όχι την περιαγωγή. Εκεί νομίζω ότι υπήρξαν οι μεγαλύτερες διαφωνίες. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία. Είναι πολλέ οι που δεν καλύφθηκαν πλήρως όπως τα θέλαμε και με ένα μέρος της συζήτησης να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα του εξαμήνου, ε, λογικό σε ένα άλλο μέρος έδωσε προσοχή και αυτό μας, ε, δεν μας κάνει εντύπωση, έδωσε προσοχή από πολιτικές δυνάμεις άλλων χωρών και άλλων παρατάξεων στα αρνητικά σημεία. Δεύτερη παρατήρηση. Η συζήτηση αυτή, όπως συχνά συμβαίνει, επικεντρώθηκε και στη χώρα προέλευσης της προεδρία. Ευκαιρία είναι το τέρμα μιας Προεδρίας, ε, η λήξη ενό εξαμήνου, είναι ευκαιρία να γίνει και μια πολιτική συζήτηση. Γίνεται πιο πολύπλοκο το θέμα βέβαια για την Ιταλία, διότι ήταν δύσκολη η μετάβαση της Ιταλίας. Διαδέχτηκε ε, μάλλον ανέλαβε σε μια φάση αλλαγής κυβερνήσεων και ε, εθνικών και πολλές φορές ε, σε συνασπισμούς κυβερνήσεων με τους οποίους έπρεπε να συνομιλήσει που συναποτελούνται από διαφορετικές πολιτικές συνιστώσεις. Περίεργο όμως βρίσκω οι Ιταλοί βουλευτές που εκπροσωπούν τη χώρα μας να επικεντρώνονται με τέτοια επιμέλεια μόνο στις αρνητικές πτυχές της χώρας μας. Και το λέω σε εσά κύριε Ταγιάννη, γιατί έχετε εργαστεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπό άλλη ιδιότητα, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε ακόμη και αν προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Λόγω χάρη ο κ. Μαλτέζε, που τώρα δεν είναι στην αίθουσα, λέει ότι η Ιταλία είναι το τρίτο κρατικό χρέο στον κόσμο. Ε, εντάξει, όντω, όντω. Το χρέος μας είναι τεράστιο. Δύο, τρει ευρώ. Όμως κανείς δεν υπογραμμίζει ότι η Ιταλία είναι πρώτη στις ε, εξοικονομήσεις, στις αποταμιεύσεις στον κόσμο. 4-3 ευρώ. Και όταν ε, οι βουλευτές από το κίνημα των πέντε αστέρων ε, μιλούν για τη φτώχεια των οικογενειών στην Ιταλία, αντιφάσκουν με τα στοιχεία τα αριθμητικά. Σε φάση κρίσης οι Ιταλικές οικογένειες είδαν να αυξάνονται οι αποταμιεύσεις τους από 3 ευρώ σε 3,9 από το 2000 2012 στο 2014. Γιατί συνέβη αυτό. Συνέβη γιατί η Ιταλική οικονομία θα μου επιτρέψει το Κοινοβούλιο που αναγκάζομαι να απαντήσω και σε θέματα εθνικά. Η Ιταλική οικονομία είναι σε φάση τρόμου, σε φάση ανησυχίας. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι μηνύματα που ε, έχουν, ε, οφείλονται όχι μόνο στη λιτότητα, που είναι μια φιλοσοφική και πολιτιστική συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε σε άλλη φάση, αλλά στον φόβο για το μέλλον. Να θεωρούμε το μέλλον ως απειλή. Τώρα, αυτούς τους μήνες, η Ιταλία ε, είδε αύξηση των αποταμιεύσεων. Οι, οι, οι οικογένειες περιέργως πλουτίζουν. Πλουτίζουν γιατί ανησυχούν και φοβούνται. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να σας πείσω για την πραγματικότητα. Όμως η πραγματικότητα λίγο-λίγο επιβάλλει την ύπαρξή της. Το λέω, το λέω σε εσά, του βουλευτέ του κινήματο των Πέντε Αστέρων που μιλάτε για τα σοβαρά προβλήματα διαφορά στην Ιταλία. Ε, το 2014 η Ιταλική Βουλή, βάσει πρόταση τη κυβέρνηση, επέλεξε, και σκεφτείτε το λίγο, ίσω δεν το έκανε αμέσω, αλλά επέλεξε ομοφόνο μετά από πρόταση τη κυβέρνηση να αναθέσει ε, την σύσταση αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς που θα διερευνήσει και την περίπτωση Μόζε, το ανέφερε η κυρία Μόη που θα επιτρέψει στη Διεθνή Έκθεση να κλείσει την εποχή ε, της παρανομίας και να ασχοληθεί πλέον με την ουσία που θα επιτρέψει να έχουμε μια νομοθεσία άνευ προηγουμένου στην Ευρώπη. Δύσκολο να επενέσει κανείς τις θετικές πτυχές της χώρας του. Γιατί εάν σκεφτεί κανείς ότι το ευρωπαϊκό βήμα είναι η ευκαιρία να μιλήσει κανείς άσχημα για τον εαυτό του, ναι, το λέω και στον κύριο Σαλβίνη, στον οποίο αναγνωρίζω συνοχή και στάση συνεπή. Όμως, πολύ καλά ε, ε, υπογράμισε τη δυσκολία και την πικρία που ε, αισθάνθηκαν οι πολίτες βλέποντας την αίθουσα του Κοινοβουλίου κενή. Όμως εγώ χαίρομαι ε, ιδιαίτερος που έμεινε στο εδρανό του κ. Σαλβίνη εξασφαλίζοντας και την ε, μεγάλη παρουσία των Ιταλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εδώ υπηρετείτε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εδώ και 11 χρόνια και είσαστε και επενδυμένοι σε ένα εθνικό αγώνα που τον σέβομαι. Όμω θα έρθετε στην προεκλογική εκστρατεία σε 3-4 χρόνια. Τρία-τρία, μην ε, δώσω μεγαλύτερη θητεία στην κυβέρνησή μα. Αλλά όταν θα έρθετε στην προεκλογική εκστρατεία θα είναι εύκολο οι πολίτε τη Ιταλία να σα πούν Εντάξει, θα ρωτήσουμε το Ρέντσι τι έκανε στην Ιταλία, αλλά εμεί θα σα ρωτήσουμε τι κάνατε κατά 15 χρόνια στην υπηρεσία τη Ευρώπη. Ε, Ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω ε, ε, εδώ κάπως πιο σύντομα στην σημερινή μας συζήτηση η πολιτική μας ομάδα που είναι ένα πρότυπο για τον κύριο η πολιτική σας ομάδα που είναι πρότυπο τον κύριο Σαλβίνη πρότεινε την αναστολή της συμφωνίας του Σέγγεν πρόκειται για ένα στόχο που η πρόεδρος Λεπέν έχει παρουσιάσει όχι εδώ στην Ολομέλεια αλλά σε συνέντευξη τύπου. Να πω τι είχε πει ο Υπουργό Εσωτερικών τη Ιταλία που συμμετείχε στο ίδιο κόμμα, την Λίγκα του Βορρά, όπου συμμετέχει και ο κ. Σαλβίνη. Να αναστείλουμε το Σέγγεν, είναι το τέλο τη Ευρώπη. Θεωρώ, έλεγε ο Μαρόνι τότε, ότι η Ιταλία θα πρέπει να αντιταχθεί πλήρω στο ε, κλείσιμο την πάυση του χώρου Σέγγεν. Αυτό ήταν το σχόλιο, ε, η παρατήρηση ε, του κυρίου Σαλβίνη που προσπαθεί να ε, αυτομολύσει προς αριστερά, αλλά δεν θα τα καταφέρει αυτά που θέλει από πολιτικής άποψης. Είναι λοιπόν πολύ απλό αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει εντυπωσιακή απόσταση μεταξύ δημαγωγίας, λαϊκισμού και πραγματικότητας. Υπάρχει μια απίστευτη απόσταση για όσους επενδύουν με συγχωρείτε, αλλά θέλω ησυχία από την αίθουσα. Ε, μου φαίνεται λοιπόν απίστευτο ως, για όσους χρησιμοποιούν πολιτικά ψευδή επιχειρήματα και ε, χρησιμοποιούν ως όπλο το φόβο για να πετύχουν τα πολιτικά τους αποτελέσματα. Και να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι σήμερα στην Ιταλία έχουμε ένα ντέρμπι. Ντέρμπι μεταξύ όσων βλέπουν τις δυσκολίες αλλά υψώνουν το ανάστημά τους και τα αντιμετωπίζουν. Προσπαθούν, προσπαθήσουμε να φανταστούμε για τη χώρα μας ένα μέλλον ε, ανάλογο της ιστορίας που μας ε, χαρακτηρίζει. Γιατί είναι πολύ εύκολο να δώσει κανείς το βάρος στην αποτυχία, στο φόβο, στο ότι τίποτε δεν θα πάει καλά. Αλλά το μήνυμα αυτό μπορεί να βολεύει προεκλογικά. Ε, να το πω και στους συναδέλφους του UKIP που δεν είναι τώρα στην αίθουσα. Πήραν προηγουμένως όμως το λόγο λέγοντας ότι εγώ χαρακτήρισα... Ε, άξες τους, τους ε, ψηφοφόρους τους. Όχι, 11 ε, εκατομμύρια ακόμα δύο όμως πολίτες δεν μπορεί να είναι ε, άνευ ευφίας. Αυτοί που είναι άνευ είναι αυτοί που δεν βλέπουν τα πραγματικά γεγονότα. Και η πραγματικότητα είναι ότι θα ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. Και θα ξεφύγουμε όχι επενδύοντας στο φόβο, όχι δίνοντας έμφαση στην αποτυχία, αλλά προσπαθώντας να κάνουμε κατανοητό ότι η μόνη δυνατή λύση για τα παιδιά μας είναι στην Ευρώπη να μην η Ευρώπη να μην είναι ένας κενός χώρος με υποσχέσεις και ωραία λόγια. Αλλά η Ευρώπη να αποκτήσει νόημα μόνο εάν στο επίκεντρο μπει η ζωή των ανθρώπων των ανθρώπων που πιστεύουν στο αύριο. Θέλουν να πιστέψουν στο αύριο, δεν φοβούνται και δεν τους νοιάζει να θεωρήσουν ό,τι συμβαίνει στον κόσμο ως απειλή. Ναι, υπάρχει στιγμία και φόβος, όμως ελπίζω ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε στην Ευρώπη να υπερισχύσουν από τους φόβους και τις απειλές οι αξίες μας. Οι αξίες που είναι τα θεμέλια της ύπαρξής μας. Αυτή είναι η διαφορά μας μεταξύ ημών και όσων ζουν στο φόβο και χωρίς γνώση. Το μέλλον που μας περιμένει εξαρτάται από την αφοσίωση του καθενός. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με την ιστορία μας, το μέλλον αυτό είναι ένα μέλλον που θα ακολουθήσει την πορεία που δείχνουν τα αστέρια της Ευρώπης. Δρόμος για την Ήπειρο και για τη χώρα μας. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ιταλική Προεδρία για τη δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Καλή τύχη στην Ιταλία, χώρα της οποίας έχω την τιμή να είμαι πολίτης. Ιδρύτρια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα λόγο στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής του τον Ζαν Κλοντ Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα για άλλη μια φορά να αποτίσω το φόρο τιμής στην τελική κυβέρνηση για την ποιότητα της δουλειάς της, στην Προεδρία και τον Προεδρεύοντα και Πρωθυπουργό κύριο Ρέντσι. Κατά τα άλλα δεν θέλω να παρατείνω την Ιταλο-Ιταλική συζήτηση. Εδώ βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν δεν απατώμε. Όπως λοιπόν και την προηγούμενη τις ε, προάλλες είχατε υποσχεθεί ότι δεν θα αναμειγνύεστε ποτέ στην εσωτερική πολιτική άλλων κρατών, σοπαίνω κι εγώ αμέσως. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Γιούγκερ. Η συζήτηση ολοκληρώνεται.